Prajem vám príjemné popoludne, dámy a páni. Budem hovoriť po slovensky, takže vás poprosím. Καλησπέρα σα. Σε Παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σα, γιατί θα μιλήσω στην μετρική μου γλώσσα. Και θα συζητήσουμε σήμερα ένα πολύ επίκαιρο θέμα την έκθεση που αφορά την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των γυναικών που ζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλα μας τα κρατημέλη έχουμε πιστεύω να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και το συζητάμε καθώς έχει να κάνει με την κατάσταση γυναικών που βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους και είμαι βεβαία πως πολλοί από εμά είχαμε και εμπειρία από πρώτο χέρι με τις γυναίκες αυτές. Εγώ ίδια γνωρίζω αρκετές ε, πολύ γενναίες γυναίκες και, αλλά και άντρες που καθημερινά δουλεύουν και τα απογεύματα και βράδια πηγαίνουν και βοηθάνε στους προσφυγικούς καταβλισμούς ή σε κέντρα υποδοχής και προσφέρουν τη βοήθειά τους σε αυτούς τους πρόσφυγες. Μου έχουν πει λοιπόν, έχουν διηγηθεί πολλές ιστορίες για αυτές τις γυναίκες που πολλές φορές δυσκολεύεται κανείς να τις πιστέψει. Γυναίκες και άνθρωποι που ψάχνουν να αναζητούν την ελευθερία και μια καλύτερη ζωή πολύ συχνά απειλούνται άμεσα. Ειδικά μια ιστορία ήταν πολύ συγκινητική, η ιστορία μιας νεαρής γυναίκας με το παιδί της που συνοδευόταν από έναν άνδρα. Η γυναίκα έτρεμε διαρκώς ανησυχούσε για, τη την υγεία του παιδιού, αλλά γιατί το παιδί είχε πυρετό, αλλά φοβόταν και για κάτι ακόμα. Προσπαθούσε ο άντρας που τη συνόδευε να την αναγκάσει να, τον να παντρευτεί έναν συγγενή, γιατί αυτό θα τους επέτρεπε να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και ίσως και σε άλλες μορφές βοήθειας και ίσως και η αίτηση ασύλου τους να διεκπεραιωνόταν γρηγορότερα. Αναγκαζόταν λοιπόν η κοπέλα αυτή να παριστάνει πως ήταν σύζυγος του εν λόγω και αυτές οι χώρες λοιπόν όχι μόνο διώκονται στις ίδιες τους τις χώρες αλλά και σε αυτές τις τόσο επικίνδυνες διαδρομές αντιμετωπίζουν ένα σωρό κινδύνους και απειλές. Θέλουμε λοιπόν να τις βοηθήσουμε να μην είναι πλέον στόχος ε, κακομεταχείρισης και είμαι βεβαία πως οι, οι προσκεκλημένες μας που είναι ειδικέ θα μας ενημερώσουν καλύτερα. Να δώσω όμως πρώτα το λόγο στην ίδια μας την εισηγήτρια, την κυρία Χάνιμπολ, που θα μας παρουσιάσει την πρωτοβουλία της και μετά θα δώσουμε το λόγο στις ε, προσκεκλημένους μας. Κυρία Χάνιμπολ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε σήμερα εδώ, πέμπτη απόγευμα, για να συμμετέχετε σε αυτή την ακρόαση. Όπως ήδη ακούσατε, θα ξεκινήσω παρουσιάζοντας την έκθεση για την οποία είμαι εισηγήτρια, που καλείται «Κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των γυναικών που ζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Όπως ήδη υπόθηκε, εδώ έχουμε συγκεντρώσει ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων που θα σας ε, μιλήσουν. Μόλις θα έχω εγώ κλείσει τη δική μου παρουσίαση, έχουν φτιάξει PowerPoint και θα αναφέρω ένα σωρό σημαντικά ζητήματα τα οποία στη συνέχεια θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Φαίνεται όντως πως κάθε εβδομάδα υπάρχουν νέες εξελίξεις και μια νέα ανακοίνωση, για μια νέα έκκληση για δράση ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση των προσφύγων. Είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά η σημερινή έκθεση είναι πολύ επίκαιρη για τις γυναίκες, γιατί η κατάσταση των γυναικών προσφυγών και των γυναικών που ζητούν άσυλο έχει παραμεληθεί μέχρι τώρα και η έκθεση προσπαθεί αυτό, αυτό να το διορθώσει. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να καλύψουμε τα πάντα σε μια μόνο έκθεση, ιδιαίτερα επειδή έχουμε περιορισμό στον αριθμό λέξεων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για κάθε έκθεση. Και έκτοτε έχουν υπάρξει εξελίξει. Το περασμένο Σαββατοκύριακο μόλις συνήφθη μια νέα συμφωνία με την Τουρκία. Αλλά εγώ στην έκθεση προσπαθώ να εστιάσω σε αυτά που θεωρώ είναι τα θέματα κλειδιά που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες και οι ετούντε άσυλα στην Ευρώπη. Και προσπαθώ ε, στη διάρκεια τη σύνταξη αυτή τη έκθεση να έρθω σε επαφή με διάφορου ε, φορεί από διάφορε οργανώσει και να ακούσω και τις εμπειρίες των ίδιων των γυναικών προσφύγων και να τις προβάλλω. Τα στοιχεία μας λένε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι περίπου το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού προσφύγων. Οι στατιστικές που αφορούν τη δημογραφική ποικιλομορφία των προσφύγων είναι δύσκολο να καταρτιστούν, αλλά γνωρίζουμε ότι περισσότεροι άνδρες φτάνουν στην Ένωση από ότι γυναίκες και παιδιά. Και αυτό νομίζω πως ε, σημαίνει πως οι άνδρες που φτάνουν εδώ δεν είναι πραγματικά πρόσφυγες και δεν θα έπρεπε όλοι να προστατευτούν διεθνώς. Αυτό το έχουμε ακούσει μάλιστα περισσότερο πρόσφατα. Αλλά ένας λόγος για τον οποίο υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ άνδρων και γυναικών είναι ότι υπάρχουν πολλοί φραγμοί για τις γυναίκες ώστε να έχουν πρόσβαση στην προστασία ε, στη διάρκεια της διαδρομής που κάνουν ή μπορεί να ξεκινήσουν. Γιατί πολύ συχνά πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά και τους ηλικιωμένους της οικογένειας. Πολλές δεν είναι ανεξάρτητες οικονομικά και γενικά στη ζωή τους ώστε να φύγουν από τη χώρα προέλευσής τους καταρχάς και όλα και περισσότερες γυναίκες που όντως φεύγουν είναι πολύ ευάλωτες σε όλα τα στάδια της διαδρομής συχνά είναι νέες, ασυνόδευτες, έγκυες ή με παιδιά αλλά και γυναίκες με ε, αναπηρίες. Μάλιστα ανακαλύψαμε ότι η βία που οφείλεται στο φύλλο είναι συχνά ο λόγος για τον οποίο οι γυναίκες φεύγουν από τη χώρα προέλευσής τους και δυστυχώς και είναι τραγικό αυτό η βία είναι και κοινή, αρκετά συχνή εμπειρία για τις γυναίκες που βρίσκονται στον δρόμο ως πρόσφυγες. Ε, ε, ακολουθούν ε, μεταναστευτικές διαδρομές και αυτό σημαίνει συγκεκριμένα προβλήματα. Όταν οι γυναίκες και οι οικογένειές τους δεν έχουν άλλη επιλογή αλλά να, από το να ακολουθήσουν επικίνδυνους δρόμους, εκτίθενται στη βία από τους εγκληματίες διακινητές. Και έχω ακούσει φρικτές ιστορίες διακινητών που εκμεταλλεύονται σεξουαλικά τις γυναίκες ως όρο για να τους προσφέρουν ε, μια θέση σε μια βάρκα που θα τις περάσει τα σύνορα. Γι' αυτό το λόγο η ασφάλεια και ε, ε, ε, μπορεί μόνο να είναι εξασφαλισμένη μέσω διάθεσης ασφαλών διαδρομών για τις γυναίκες που φεύγουν από διώξεις στις χώρες τους. Οι πολιτικές ασύλου πολύ συχνά παραβλέπουν την ειδική θέση των γυναικών που αναζητούν άσυλο και πολύ συχνά εξετάζονται μόνο υπό το φως των ανδρικών, της ανδρικής εμπειρίας. Παρά το ότι έχουμε κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές στα κράτη-μέλη και οι διαφορές είναι αρκετά σημαντικές. Υπάρχει μάλιστα μεγάλο χάσμα στην προστασία που προσφέρεται στις γυναίκες που αναζητούν άσυλο στην Ένωση. Καταρχήν θα ήθελα να σας ε, μιλήσω για το πώς αντιμετωπίζετε το φύλλο στην λήψη της απόφασης το ποιος θα πάρει το καθεστώς ασύλου, ε, πρόσφυγα συγγνώμη, και ποιος όχι. Υπάρχουν συγκεκριμένες ε, κατευθύνσεις γραμμές για το φύλλο, αλλά δεν είναι δεσμευτικές και αποτελεσματικότητά τους ήταν μερική και άνηση. Και εγώ σίγουρα είμαι υπέρ ενό νέου συνόλου ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραμμών. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι βλάβες που στις οποίες υπόκειται οι γυναίκες ε, λόγω του, είναι, του ότι είναι πρόσφυγες πολύ συχνά προκαλούνται από συζύγους ή συντρόφους και η Διεθνής Νομοθεσία αναγνωρίζει ότι η δίωξη συμβαίνει όταν το κράτος δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να προστατέψει τις γυναίκες που βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση. Κατά συνέπεια θα πρέπει να το δούμε ε, και από την οριζόντια και από την κάθετη διάσταση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο το, της γενετήσιας ε, βίας. Είναι σαφές ότι πολλά κράτη-μέλη, 12 μάλιστα, δεν έχουν ακόμα υπογράψει ούτε κυρώσει τη σύμβαση της ε, Ισταμπούλου. Και όπως γνωρίζετε, αυτή η σύμβαση επιβάλλει στα κρατη... απαιτεί από τα κρατημέλη να ερμηνεύουν την αίτηση, το καθεστώς πρόσφυγα ε, με βάση το φύλλο, καθώς και να παρέχουν εκθέσεις σχετικές με το φύλλο στην εξέταση της καθέτησης. Την περασμένη εβδομάδα ήταν η Παγκόσμια ημέρα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Λόγω της φύσης ε, όμως ε, της κατάστασης είναι πολύ λιγότερο πιθανόν οι γυναίκες να έχουν ε, τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι προφορικές μαρτυρίες πολλές φορές παίζουν ρόλο, ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιολόγηση αξιοπιστίας. Όταν οι γυναίκες έχουν υποστεί τραύμα μπορεί να είναι απρόθυμες ή να αποκαλύπτουν πολύ αργά τις σχετικές πληροφορίες και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Έκουσα από ΜΚΟ και από πρόσφυγες γυναίκες που μιλούν για την, την οτροπία της δυσπιστίας, ότι δηλαδή οι αρχές δεν τις πιστεύουν εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι δεν καταφέρουμε να λάβουμε υπόψη την περιπλοκότητα των αναμνήσεων, της βλάβης και του τραύματος και ότι επιβαρύνουμε πάρα πολύ τις γυναίκες πρόσφυγες που ζητούν άσυλο. Θα πρέπει λοιπόν να καταρτιστεί καλύτερα το προσωπικό. Ακούσαμε πολλές ε, νέες προτάσεις πρόσφατα από την Κομισιόν ως τμήμα της ατζέντα για τη μετανάστευση και την ανταπόκριση στη κρίση την προσφυγική. Και εγώ θα ήθελα να, πω, να μιλήσω για μια πρόταση συγκεκριμένα, την πρόταση για ένα κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών προέλευσης. Αυτός ο προτινόμενος κανονισμός ε, θίγει πολύ σημαντικά θέματα όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών που ζητούν άσυλο στην Ένωση. Καμιά χώρα δεν μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλής για τις γυναίκες και για τα κορίτσια όταν η βία λόγω φύλου, η γενετήσια βία είναι μια πανδημία. Δεν υπάρχουν ε, κανόνες και πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση ανάμεσα στην κατάσταση των γυναικών και των ανδρών. Τώρα, αν στραφούμε στις γυναίκες και στις ανάγκες των γυναικών που βρίσκονται σε διαδικασία αίτησης ασύλου, υπάρχουν ε, και εκεί διάφορα περίπλοκα στοιχεία. Καταρχήν, οι γυναίκες αυτές χρειάζονται πρόσβαση στην νομική συμβουλή. Όμως ε, τα ψυχολογικά τραύμα, η ντροπή, και ο στιγματισμός ε, λόγω της βίας μπορεί να καταστήσουν δύσκολο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους οι, οι, δικηγόροι ή οι σύμβουλοι. Είναι απαραίτητο λοιπόν η γυναίκα να, έχει τη δυνατο... την... να κερδίσει την να... να εμπιστευτεί τον σύμβουλο ώστε να του αποκαλύψει λεπτομέρειες. Ε, Ενώ οι περικοπές στην ε, νομική αρρωγή είναι πραγματικότητα στα περισσότερα κράτη-μέλη. Πολλές γυναίκες λοιπόν μένουν χωρίς καμιά άλλη επιλογή. Παρουσιάζονται μόνες τους ε, στις ε, διάφορες ακροαματικές διαδικασίες. Και είχα τέτοιου είδους εμπειρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ορισμένες από τις συστάσεις που θα υποβάλω με την έκθεσή μου περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζητά κανείς γυναίκα, διερμηνέα και ε, συνομιλητή. Επίσης ε, να μπορεί να μιλήσει έτσι πιο εύκολα για το τραύμα, την σεξουαλική βία ενώ οι ε, τροπολογίες ε, ε, μιλούν για τις συνθήκες υποδοχής και πολλά προβλήματα υπάρχουν εκεί και αυτά είναι η κατάρτιση ειδικά με βάση το φύλλο για το προσωπικό που εργάζεται εκεί και η καθολική ενημέρωση όσον αφορά την σεξουαλική βία και τον κροτηριασμό των γυναικείων οργάνων. Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ε, προγεννητική υγεία, ε, και ούτω καθεξής. Είμαι πολύ σαφή στην έκθεσή μου ότι η κράτηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως τελευταία ίστατη λύση. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τους ε, επιβιώσαντες σεξουαλικής βίας και τις έγκυες γυναίκες. Πολύ συχνά παραβλέπετε ότι ότι οι γυναίκες μπορεί να υποφέρουν από βία και από τη στιγμή που βρίσκονται πια στην Ένωση. Πολύ συχνά από, υπόκειται βία από τους ίδιους τους συντρόφους τους και δυστυχώς και από το προσωπικό που τις υποδέχεται και από αυτού θα πρέπει άμεσα να δενεργήσει και να δράσει η Ένωση. Τέλος, να πω δύο λόγια για την ένταξη. Οι γυναίκε πρόσφυγε αντιμετωπίζουν ειδικέ προκλήσει, ιδιαίτερε προκλήσει όσον αφορά την ενταξία του και συχνά είναι αντικείμενο διακρίσεων. Ε, έτσι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, βία και φτώχεια. Πολλέ από τι γυναίκε που ζητούν άσυλο ζουν κάτω από το όριο τη φτώχεια, συμπεριλαμβανομένων των εγγύων και των νεαρών μητέρων. Ακόμα και όταν του έχει χορηγηθεί το καθεστώ ασύλου, πολύ συχνά συναντούν σημαντικά εμπόδια για να βρουν απασχόληση. Η φροντίδα των παιδιών είναι πολύ σημαντική εδώ και γι' αυτό και προτείνω τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν καλύτερα και ε, περισσότερο το Ταμείο Συνοχής πέρα από το Ταμείο Ασύλου και ε, ένταξη, ώστε να προωθηθεί η ένταξη αυτών των γυναικών στην αγορά εργασία. Η φροντίδα των παιδιών είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουν ε, οι γυναίκε πρόσφυγε να ενταχθούν στην κοινωνία και θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στην επίγουσα κατάσταση την ανθρωπιστική στην Ευρώπη και στις γειτονικές της χώρες, αλλά πρέπει τώρα να ε, σχεδιάσουμε όλα αυτά ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την επιτυχή ένταξη αυτών των ανθρώπων. Όμω πολύ είναι είναι οι στατιστικές οι πρόσφατες. Μετά από τι φρικτέ επιθέσει στο Παρίσι, τον περασμένο εβδομάδα 300 επιθέσεις ρατσιστικού τύπου έγιναν στο Λονδίνο και πολλέ από αυτέ τι επιθέσει ήταν κατά γυναικών. Τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να προωθήσουν τη δημιουργία ενό ασφαλού ευνοϊκού περιβάλλοντος και να τα πολεμήσουν κάθε είδος διάκριση. Διανύουμε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση. Η ανταπόκρισή μας στην μετανάστευση και στην των προσφύγων θα πρέπει να συνδυάσει μέτρα ώστε να ελαφρυνθεί ε, το πρόβλημα με πιο μακροπρόθεσμες λύσεις. Η τεράστια ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη φυσικά μας ανησυχεί οι άνεσε σχέσεις ε, μεταξύ των φίλων μεγιστοποιούνται στη διάρκεια μιας κρίσης και αναπόφευκτα οι καιροί κρίσεις καθιστούν τις σχέσεις μεταξύ των φίλων πιο δυσχερείς. Η πίεση δε στις χώρες που αντιμετωπίζουν το προσφυγικό δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο να μην προστατευτούν όπως πρέπει οι γυναίκες. Πρέπει να βλέπουμε πιο μακροπρόθεσμα. Αυτή η φάση αβεβαιότητα παρουσιάζει, είναι ταυτόχρονα μια ευκαιρία ώστε να δημιουργηθούν πιο διάσημες πολιτικές που θα λειτουργήσουν καλύτερα στο μέλλον. Πρέπει να είμαστε πιο ανθεκτικοί, να σκεφτούμε πιο στρατηγικά για να προστατεύσουμε τις γυναίκες και τους, και, που ζητούν άσυλο και τι πρόσφυγες στο μέλλον. Το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να εξαφανιστεί τώρα κοντά. Ιδιαίτερα ο πληθυσμό τη Ευρώπη που γερνά και η δημογραφική πρόκληση που σημαίνει αυτό, ενώ θα έπρεπε να επεκτείνεται ο πληθυσμό μα, θα έπρεπε να μα οδηγήσει στο να υποδεχτούμε, ε, να καλωσορίσουμε μάλιστα τους πρόσφυγε και να σκεφτούμε πόσο καλό και πόσο θετική θα είναι η συμβολή των γυναικών στις κοινωνίες μας. Η έκθεση αυτή είναι μια ευκαιρία για να σχηματίσουμε, να, να δρομολογήσουμε την προσέγγιση προς το άσυλο έτσι όπως την επιθυμούμε εμείς. Σας ευχαριστώ κυρία Χάνιμπολ για την ε, θαυμάσια αυτή και ιδιαίτερα περιεκτική και περίπλοκη έκθεση που δεν αρκείται μόνο να περιγράψει τι πρέπει να πράξουμε υπέρ των γυναικών που προσέρχονται και χρειάζεται τη βοήθειά μας, αλλά δείχνει και ότι στις χώρες μέλη δεν πρέπει να κυριαρχήσει ο, φόρο, ο φόβος συγγνώμη, και η απόρριψη απέναντι στους ε, πρόσφυγες. Θα δώσω το λόγο τώρα στις εμπειρογνώμονες που προέρχονται από διάφορους θεσμούς Πρώτη την κυρία Ανδρέα Βόνκεμαν από τον ύπατο αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Θα μιλήσει για γυναίκες και κορίτσια και τα δεινά που υφίστανται καθώς προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Thank you, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία που δίνετε στον ύπατο αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών να σας μιλήσει για την ανάγκη προστασίας γυναικών και κοριτσιών σε αυτές τις έκτακτες περιστάσεις. Έχουμε διαβάσει την έκθεση πρωτοβουλία της κυρίας Χάνιμπολ με μεγάλο ενδιαφέρον. Στηρίζουμε την ανάλυση της για τα κενά που ε, υπάρχουν καθώς και τις συστάσεις που κάνει. Ως τώρα 2015 πάνω από 800.000 άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη από τη θάλασσα, 730.000 από την Ελλάδα και 150.000 περίπου ε, στην Ιταλία. 34% των προσώπων αυτών είναι γυναίκες και παιδιά. Εκτός από τους κινδύνους και ε, τις προσβολές και, όσα άλλα υφίστανται στη διάρκεια του ταξιδιού τους για να φτάσουν στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουν κινδύνους και στην κίνησή τους μέχρι να φτάσουν στα, παρά, στα παρά, παράκτης περιοχές της Ευρώπης. Αυτές είναι και οι οδοί που χρησιμοποιούν, οι διαδρομές καλύτερα που χρησιμοποιούν να βλέπετε στο χάρτη, στη διαφάνεια είναι οι διαδρομές που ακολουθούν συνήθως οι ε, πρόσφυγες με τα σημεία συναντοπίζονται στα σύνορα μεταξύ ε, Ελλάδος και Φιρόμ καθώς και Φιρόμ και Σερβίας, Σλοβενίας και Κροατίας μπορεί να αλλάξουν οι διαδρομές αυτές τώρα και να περάσουν από άλλες χώρες. Στο μεταξύ πάντως άνθρωποι που δεν είναι ε, από Συρία, Ιράκ ή Αφγανιστάν έχουν κολλήσει στα σύνορα και είναι γνωστή τώρα η κατάσταση που διαμορφώνεται στα ε, σύνορα Ελλάδας-Μακεδονίας ε, όπου γυναίκες και παιδιά αναγκάζονται να διαγνυκτερεύουν σε εντελώς ακατάλληλα και ανασφαλή μέρη. Ορισμένοι έχουν επιστρέψει στις Αθήνες, ορισμένες έχουν επιστρέψει στις Αθήνες, στην Αθήνα δηλαδή, ε, με λεωφορεία που διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση. Άλλοι φαίνεται να χάνονται, να εξαφανίζονται από την περιοχή των συνόρων. Παρ' όλα αυτά, οι εντάσεις ανάμεσα σε αυτούς και αυτές που παραμένουν μετά στα σύνορα αυξάνουν. Στον πίνακα βλέπετε, κάποιες στατιστικές, βλέπετε μια εχμή αφήξεων τον Οκτώβρη. Βλέπουμε τώρα να μειώνονται κάπως οι αριθμοί, ίσως λόγω και των συζητήσεων που διεξάγονται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Τουρκίας ίσως και λόγω των συνθήκων, ίσως και λόγω άλλων άγνωστων ε, ε, αιτιών. Πρώτα λοιπόν ε, Σύριοι, Αφγανοί, Πακιστανοί και Ιρακινοί και Ιρακινές εννοείται φτάνουν στην Ελλάδα, στην Ιταλία, τα πράγματα είναι διαφορετικά σε ό,τι αφορά τι εθνικότητες, κυρίως προέρχονται από Ερυθρέα, Νιγηρία, Σομαλία και Σουδάν. Οι γυναίκες δεν είναι καθεαυτές ευάλωτες. Οι γυναίκες, μάλλον είναι καθεαυτές ευάλωτες. Και εφόσον δεν συνοδεύονται από άνδρες συγγενείς, είναι ακόμα πιο ευάλωτες. Αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εκμετάλλευσης, ε, ε, γενετήσιας βίας και ούτω καθεξής. Αντιμετωπίζουν κινδύνους και σε ε, εγκαταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ φορτωμένες, είναι επίσης ε, ευάλωτες σε ε, επιθέσεις και άλλους κινδύνους σε σημεία όπου παίρνουν λεωφορεία κλπ. ή σε σημεία transit ή σε καταλήμματα εφόσον αυτά είναι αβέβαια και χωρίς προστασία. Ο ύπατος αρμοστής έχει παρουσία σε όλες τις ε, χώρες από τις οποίες περνούν οι πρόσφυγες. Έχουμε ακούσει αναφορές για γυναίκες και παιδιά, μεταξύ αυτών και αγόρια, που αναγκάζονται να πληρώσουν τους διακινητές με ε, σεξουαλικές υπηρεσίες, το για να μπορέσουν να περάσουν, για να φτάσουν στην χώρα προορισμού. Γι' αυτό ο ύπατος αρμοστής των Ενωμένων Εθνών για, τις, για τις πρόσφυγες και η UNPA έχουν αναλάβει να χαρτογραφήσουν τα προβλήματα αυτά στις χώρες της Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων και θα σας μιλήσω και για τα βασικά αρχικά συμπεράσματα των αναφορών αυτών σε λίγο. Άλλο ε, που σημειώσαμε από την κρίση αυτή είναι τα πολύ νεαρά κορίτσια που εξανακάζονται σε γάμο και από την Συρία αλλά και σε χώρες προορισμού, στην Ευρώπη. Ακούσαμε ιστορίες και από υπηρεσίες της χώρες προορισμού ότι τα κορίτσια αυτά στέλνονται από τους γονείς τους με την ελπίδα ότι θα είναι ασφαλής εφόσον ή συνοδεύονται από συγγενή ή φτάνουν και μόνες τους στην Ευρώπη όπου θα εξαναγκαστούν σε γάμο με κάποιον ο οποίος είναι ήδη εγκατεστημένος στην Ευρώπη. Αυτό βεβαίως είναι πηγή μεγάλης ανησυχίας και πρέπει να εξεταστεί. Διότι βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ανήλικα κορίτσια, πολύ κάτω από το όριο ηλικίας για γάμο και δεν είναι βέβαια για το καλό του παιδιού να εξαναγκαστεί σε τέτοιο γάμο. Επίσης, χωρισμός από την υπόλοιπη οικογένεια είναι μέγα θέμα σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γίνεται σε σημεία εισόδου, εξόδου. Οι υπηρεσίες του ΥΠΑ του Αρμοστού εργάζονται πραγματικά ε, χωρίς ε, σταματημό για να αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα χωρισμού οικογενειών και για να μπορέσουν να επανενώσουν τις οικογένειες επιτόπου μόλις ε, ε, ε στην υπόψη τους ένα τέτοιο γεγονός. Άλλη μεγάλη πρόκληση και άνευ προηγουμένου για τον ύπατο αρμοστή είναι ότι ευάλωτοι άνθρωποι και γενικά οι άνθρωποι ε, δεν θέλουν να αναγνωριστούν ως ευάλωτοι γιατί και αυτό είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις έχετε λοιπόν ε, γυναίκες μοναχές τους ε, ασυνόδευτα ανήλικα τα οποία διακινούνται και λένε αχ, αυτό να, αυτός είναι ο συγγενής μου», για να μην φανεί ότι είναι μόνα τους. Και αυτό βέβαια γίνεται και αντικείμενο κατάχρησης. Είναι τόσο, έχουν ε, ε, τέτοια ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί να προχωρήσουν, να συνεχίσουν την πορεία αυτή προς την χώρα προορισμού, που ε, δεν θέλουν να τους ανακόψει τίποτα και θεωρούν ότι αυτό μπορεί να σταματήσει την πορεία τους. Κάτι που αναφέρει και η κυρία Χάνιμπολ στην έκθεσή της είναι τα της υποδοχής. Και αν μπορούν να τηρηθούν τα πρότυπα του κεκτημένου της Ευρώπης για την υποδοχή ε, προσφύγων κέντρα υπερφορτωμένα και στις χώρες υποδοχής με καταστάσεις όπου γυναίκες και οικογένειες δεν, είναι, δεν διαμένουν χωριστά από ε, μόνους τους ενήλικους άνδρες. Το άρθρο 18 παράγραφος 9 της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής λέει ότι εφόσον υπάρχει πίεση σε ένα ε, σύστημα υποδοχής, τότε για σύντομα διαστήματα η χώρα μέλος μπορεί να προσφέρει τις βασικές ε, υπηρεσίες σε όσους ζητούν το άσυλο. Ποιες είναι όμως αυτές οι βασικές ανάγκες. Είναι τροφή, νερό, ε, βασικές ε, υπηρεσίες υγείας. Όχι, μιλούμε εδώ και για ε, βασικές υπηρεσίες καταλήματος, δηλαδή και οι γυναίκες και τα παιδιά να μπορούν να, είναι, να διαβιούν ξεχωριστά από τους άνδρες. Τώρα για την relocation, επανεγκατάσταση. Λέει στην απόφαση του Συμβουλίου ότι θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε ευάλωτα πρόσωπα. Το ερώτημα είναι πώ θα γίνει στην πράξη με όλου αυτού του ανθρώπου που δεν θέλουν να αναγνωριστούν ότι είναι μόνοι του και άρα εδώ η πρόκληση είναι να μπορέσει να αποκαταστεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται σε, στην κίνηση έτσι ώστε να πάνε στα hot spot τα οποία ιδρύονται. Το πρόβλημα με αυτά τα hot spot είναι, όσο γνωρίζετε, ότι ακόμα καθυστερούν και ούτως ή άλλως ιδρύονται και λειτουργούν πάρα πολύ αργά. Άλλη σημαντική προϋπόθεση για τα hot spot και επανέρχομαι εδώ στο θέμα της υποδοχής είναι να είναι σωστή η υποδοχή. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Για να σας δώσω μια ιδέα, με συγχωρείτε με τη διαφάνεια μια στιγμή, για τον αριθμό θέσεων που είναι διαθέσιμες από τις 23 ενδεκάτου, 3.600 από 160.000 που χρειάζονται από ε, την Ιταλία μετεγκαταστάθηκαν 130 άνθρωποι και από την Ελλάδα 30. Αυτό απέναντι στις δεκάδες χιλιάδες που παραμένουν ακόμα εκεί. Άλλο θέμα είναι και οι ποσοστώσεις. Οι χώρες μέλη έχουν ποσοστώσεις, συχνά είναι πολύ περιοριστικές. Αυτό χρειάζεται βέβαια ταχεία διεκπαιρέωση και πρέπει να τηρήσουν τα επισημένα οι χώρες μέλη, να προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες σε γυναίκες που έχουν υποστεί ε, γενετήσεις επιθέσεις κ.ο.κ. Αναφερθήκατε πριν και στην εθνικότητα. Ανεξαρτήτως εθνικότητας δεν πρέπει να, διακρίνονται, να γίνονται διακρίσεις σε βάρος των γυναικών που έχουν ε, υποστεί επιθέσεις κ.ο.κ. Και εδώ Είναι βέβαια και αμφισβητήσιμη και η έννοια της ασφαλούς χώρας προελεύσεως. Το πρόβλημα επίσης είναι ότι άνθρωποι που δεν επιθυμούν να συνεργαστούν, δηλαδή πρόσφυγες που δεν επιθυμούν να συνεργαστούν, ποια είναι η καλύτερη απάντηση, κράτηση για ανθρώπους που πρόκειται επίσης να μετεγκατασταθούν, ε, πού και πώς, αυτό είναι επίσης ένα άλλο δίλημα. Και πολύ σύντομα σε ό,τι αφορά πάλι τα καταλήματα, οι γυναίκες και τα κορίτσια και ιδίω όσα βρίσκονται σε κίνδυνο θα πρέπει να έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα hot spot. Θα πρέπει να είναι επαρκή η υποδοχή ως προϋπόθεση για την έλευσή τους στα hot spot. Θα πρέπει να χορηγείται ενημέρωση για τις επιλογές και με τρόπο που να ε, συμφωνεί και με το φύλλο και με την ηλικία του προσώπου. Οι χώρες μέλη πρέπει να θυμηθούν ότι η κράτηση και τα κέντρα κράτησης πρέπει να είναι πραγματικά η στάτη καταφυγή. Και σύμφωνα και με τις κατευθυντικές γραμμές του είπα του αρμοστή, γυναίκες που είναι έγκυοι, ε, θύματα βιασμών ή θύματα βασανιστήριων δεν πρέπει καταρχήν να κρατούνται. Σε ό,τι αφορά το nationality screening, να μην γίνεται επανεισδοχή, ιδίως από χώρες όπου υπάρχει για παράδειγμα υψηλό κίνδυνος να υποστούν γενετήσεις επιθέσεις ή άλλες διώξεις στη βάση του φύλου. Ο επίσης λέει στην εκθεσή της η κυρία Χάνιμπολ ότι πρέπει να έχουν και πρόσβαση σε γυναίκες συνομιλήτριες που θα κάνουν τη συνέντευξη δηλαδή καθώς και σε γυναίκες διερμηνείς και να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες υποβολής αίτησης ασύλου και να χαίρουν διεθνούς προστασίας. Τέλος, υποστηρίζουμε αυτό που λέει στην εκθεσή της η κυρία Χάνιμπολ για περισσότερες νόμιμες διαδρομές και για τις γυναίκες με την κατάσταση ανθρωπιστικές μεταφορές, ανθρωπιστικές βίζες και ούτω καθεξής. Και μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Είναι σημαντικό λοιπόν να αντιληφθούν οι χώρες μέλη ότι εφόσον υπάρχουν αυτά τα ρυθμισμένα συστήματα θα πρέπει και θα μπορούν να ελέγχουν πολύ καλύτερα και ποιο εισέρχεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για ε, γραμμέ γραμμές ανάλογα με το φύλλο και για την χορήγηση ασύλου και τα άλλα δικαιώματά τους. Θα θέλαμε επίσης να συστήσουμε οι κατευθυντήρες αυτές γραμμές ε, να εξετάσουν βέβαια και άνδρες και γυναίκες που ενδέχεται να έχουν ε, προβλήματα σχετιζόμενα με το φύλλο. Πριν δεστρώστε κυρία Ρέλη. Να καλωσορίσω δύο ομάδε επισκεπτών από τη Σουηδία και την Ιταλία αντιστοίχως. Καλώς ήλθατε. Κύριε Ράιλι, έχετε τον λόγο. Είστε από την Επιτροπή Γυναικών Προσφύγων από τη Γενέβη. Θα μας μιλήσετε για την προστασία των γυναικών προσφύγων στην Ευρώπη. Ένα σκανδαλώδε έλλειμμα. Καλησπέρα σας. Είμαι η Rachel Riley. Εκπροσωπώ την Επιτροπή Γυναικών Προσφύγων από τη Γενέβη. Υποστηρίζουμε την βελτίωση των συνθήκων ζωής γυναικών, κοριτσιών, παιδιών που είναι θέματα εκτοπισμού. Διεξάγουμε έρευνες, δημοσιεύουμε συμπεράσματα, διατυπώνουμε προτάσεις και συστάσεις για αλλαγή. Ασχολούμεθα με ευρύ φάσμα θεμάτων από την πρόληψη της σεξουαλικής και φιλετική βίας ως την βελτίωση των συνδικών ζωή των γυναικών, πρόσβαση σε αναπαραγωγική υγεία, φροντίδα για απάτηδες και ούτω καθεξής. Ο λόγος για τον οποίο είμαι σήμερα εδώ είναι ο εξής. Η έδρα στη Γενέβη. Όμως, έχουμε αντικείμενο ανά την Ευρώπη. Παραδοσιακά αρχές Νοεμβρίου κάθε χρόνο συμμετέχουμε σε μεικτή αποστολή αξιολόγηση με την υπετερμοστία του ΟΗΕ για να διερευνήσουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν γυναίκες και παιδιά στην σημερινή κρίση. Έχουμε πείρα ως ε, θεσμός και προτείνουμε μέτρα προστασίας για γυναίκες και παιδιά. Και για γυναίκες και κορίτσια, με συγχωρείτε. Εξετάσαμε την κατάσταση στην Ελλάδα. Πήγαμε στην Αθήνα και σε δύο νησιά, στη Χίο και στην Σάμο, στην Ελλάδα, παραλαμβάνω, που αφήγνεται πρόσφυγε, πήγαμε στα Σκόπια στην πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, στη Γεβιελή, στα σύνορα Μακεδονία Ελλάδο και όσο το πενόψε στα σύνορα Μακεδονία Σερβία. Όπω είπε η κυρία Χάνιμπολ και όπω είπε και η συνάδελφο από την Ερμοστία, πρόκειται για κρίση προσφύγων χωρί προηγούμενο. Το πλήθο μεταναστών και προσφύγων που ταξιδεύουν ταχύτερα διερχόμενοι από διάφορες χώρες, καθιστά την κατάσταση πολύ διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν. Είναι μια διαφορετική κρίση προσφύγων, η οποία απαιτεί μια συντονισμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Διότι όλοι αυτοί φοβούνται ότι θα κλείσουν τα σύνορα, το βλέπουν αυτό και φοβούνται και τον επερχόμενο χειμώνα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα του πόσο καταπιούσα είναι η κατάσταση, φανταστείτε μια γυναίκα, η οποία, είναι, ήταν 9,5 των ε, μηνών με έγκυος και η οποία δούλευε, μετανάστευσε και δεν πήγαινε καν στο μεστήριο μέχρι που την έπεισε η οικογένειά της να πάει σε μεστήριο στην Ελλάδα. Δεν είχε μόνο άλλο χρόνο, λίγες ώρες μετά τη γέννηση ξανάφυγε και συνέχισε το ταξίδι της. Όπω είπε και η συνάδελφο από την υπερδιαγνωστία, ανησυχούμε διότι καθώς κλείνουν τα σύνορα, όπως προείπα, δεν υπάρχει συντονισμένο σχέδιο αντιμετώπιση της έκτακτη ανάγκης. Ειδικά για τους μη Συρίου, οι Σύριους οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι σε διάφορα σημεία χωρίς ε, ανθρωπιστική υποστήριξη. Η κίνηση λοιπόν, η εφετηρία αν θέλετε για μας είναι η Η μεικτή λοιπόν επιτροπή, η ISC, που είναι η μεικτή επιτροπή μεταξύ Εθνών και όλων των άλλων οργανώσεων. Η επιτροπή αυτή θέσπισε κατευθυντήριε γραμμέ, σύμφωνα με τις οποίε όλο το προσωπικό ανθρωπιστικών οργανώσεων πρέπει να θεωρεί ότι συμβαίνουν περιστατικά σεξουαλικής βίας και ότι έτσι επηρεάζονται οι πληθυσμοί. Πρέπει η απειλή αυτή να αντιμετωπιστεί σοβαρά, να φέρει την απειλή τη ζωέ γυναικών και κοριτσιών, ακόμη και αν δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία. Αυτό είναι γενικά το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε απόψε. Η βία λοιπόν αυτή, αυτή η σεξουαλική βία, συμβαίνει να είναι μια πραγματικότητα και υπάρχουν πολλέ γυναίκε και κορίτσια που είναι θύματα αυτή τη βία και αυτό συμβαίνει ακόμη και αν δεν υπάρχουν απόλυτε αποδείξει σχετικά με την τέλεση αυτών των περιστατικών. Κατά τη διάρκεια των 7 ημερών διαπιστώσαμε ότι γυναίκες και κορίτσια χρήζουν καλύτερες προστασίες, υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα από την κοινωνία βεβαίω ε, και όλους τους ε, άλλους εμπλεκομένους, αλλά υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα. Συμβαίνουν μορφές βίας που θα περίμενε κανείς οικιακή βία, βιασμό, σεξουαλική βία, σεξουαλική παρενόχληση, σωματικέ επιθέσει, φυσική βία, σωματική βία και τράφικινγκ, εμπόριο ανθρώπων. Η βία αυτή κατά κύριο λόγο αφορά τις πλέον ευάλωτε ομάδες, μόνες γυναίκες που ταξιδεύουν, γυναίκες που ταξιδεύουν με παιδιά, εγγύου, ε, γυναίκες σε λοχεία, εφήβους, ασυνόδευτα παιδιά, ανυπαδρές νεαρέ γυναίκες καμιά φορά με παιδιά και αναπηρέ γυναίκε, γυναικέ με αναπηρίε. Η συνήθι αντίδραση που συλλέξαμε είναι ότι δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα οι, οι δικοί μα εντόπισαν σχεδόν αμέσω μια γυναίκα από χώρα τη Ποσοχαρία τη Αφρική, η οποία ταξίδευε μόνη τη προ Γερμανία. Έφυγε λόγω πολιτικών διωγμών στη χώρα της. Είχε φύγει πριν από ένα μήνα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της υποβλήθηκε δύο φορές σε σεξουαλική βία εδώ στο διαβατηριό της. Κοιμήθηκε έξω στην Ήπεθρο, σε ένα ελληνικό νησί, χωρίς ε, καμία προστασία, χωρίς καταφύγιο και χωρίς καμία υπηρεσία δεν κατέστη δυνατόν να καταγραφεί. Δεν είχε λάβει καμία βοήθεια κανένα είδου σε όλη αυτή την περίοδο. Τα ευρήματά μας λοιπόν δείχνουν ότι παρά τις ενδείξεις για σεξουαλική βία που υποτίθεται μόνο ενδείξεις εμείς ε, δεν είδαμε αντιθέτως καμία προσπάθεια πρόληψης αυτής της βίας. Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις όπου μένουν για λίγο οι πρόσφυγες, ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά, δεν προσφέρουν παρά τα ελάχιστα τα, βασικά. Ας πούμε σε κέντρο κράτηση ήταν καλοκαίρι. Δεν υπήρχαν καν ξεχωριστές τουαλέτες ή ντους για γυναίκες και άνδρες. Μια αερακινή η οποία έμεινε στο κέντρο μας είπε ότι πήγοντας την τουαλέτα στο ντους αισθανόταν εντελώς ανασφαλής. Ε, και εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα βασικό μέτρο, αυτός ο βασικός διαχωρισμός δηλαδή τουλάχιστον για τις εγκαταστάσεις υγιεινής. Είναι το απολύτως ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει κανείς σε γυναίκες και κορίτσια. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός για ενέργειες πρόληψης. Δεν υπάρχει ούτε καν πρόγραμμα αντιμετώπισης των περιστατικών όταν συμβαίνουν. Δεν υπάρχει ούτε καν συνεννόηση μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων. Η στάση, όπω είπα, ήταν εν γέννη ότι αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν. Δεν υπάρχει σεξουαλική βία. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολύ λίγα περιστατικά καταγγέλλονται. Και αυτό είναι ένα φαύλο κύκλο. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν συμβαίνουν τα περιστατικά. Λοιπόν, το γενικότερο επίπεδο γνώση του προβλήματο είναι πολύ χαμηλό μεταξύ των ε, οργανώσεων και γι' αυτό είναι και δύσκολο να δημιουργηθούν κατάλληλες υπηρεσίε εκεί όπου δεν υπάρχουν. Η ομάδα μα πήρε συνεντεύξεις ε, από πολλούς, ε, ξέρω μια γυναίκα με την κόρη της που είχε δώσει ένας, έναν άλλο άνδρα και ο οποίος του επιτέθηκε, τη απείλησε. Βρέθηκαν αυτές οι δύο γυναίκες σε κατάσταση κλονισμού δεν είχαν πρόσβαση κανένα είδου πληροφορία, όπως καμιά ε, συμβουλή ή αλλε υπηρεσιε Οι συστάσεις μα, οι βασικές μας τουλάχιστον συστάσει είναι για να προστατεύσουμε καλύτερα γυναίκε και κορίτσια χρειάζεται περισσότερο καλύτερο συντονισμό. Όχι απλώ ύπαρξη μια υπηρεσία στη συγκεκριμένη χώρα, αλλά και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών χωρών. Καλύτερο συντονισμό μεταξύ διεθνών, εθνικών και τοπικών οργανώσεων. Διπιστώσαμε ότι οι αντιδράσει, όποιε και είναι αυτέ, δίνονται χωρί κανένα συντονισμό. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη συνεργασία. Υπάρχουν στεγανά. Πρέπει όταν υπάρχουν περιστατικά ή ας πούμε μια γυναίκα βιαστή στην Ελλάδα πρέπει η πληροφορία αυτή σχετικά με την υπόθεσή της να μετακυληθεί στις υπηρεσίες στη χώρα στην οποία θα πάει για να μπορέσουν να την υπεριθάλψουν. Χρειάζεται λοιπόν και καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία. Επίσης, χρειαζόμαστε εκπαιδευμένο προσωπικό επιτόπου για αυτή τη μορφή βίας καλύτερο συντονισμό επίση με την κοινωνία των πολιτών, με ομάδες υποστήριξη γυναικών. Και όπω είπε και η συναδελφό μου, χρειαζόμαστε περισσότερη πρόσβαση σε γυναίκε διερμηνείς για να διευκολύνουμε τη συζήτηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλύτερα εκπαιδευμένου ειδικού επί θεμάτων σεξουαλική βία επιτόπου και εν κατακλείδη πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κατάλληλε υπηρεσίε παρέχονται στι γυναίκε. λόγω της φύσης της κρίσης και το ότι οι πληθυσμοί μετακινούνται ταχύτατα, οι σχετικές υπηρεσίε πρέπει να παρέχονται από ανθρώπους επιτόπου, μεταξύ άλλων να παρέχεται και ψυχολογική υποστήριξη. Πρέπει να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι, ασφαλείς θύλακες για γυναίκες και κορίτσια στους προορισμούς. Και εξίσου σημαντικό, χρειάζεται ο ιατρικός εξοπλισμός, ο οποίος να είναι προσβάσιμος αμέσως ιδιαίτερα σε περιπτώσει που οι άνθρωποι δεν πρόκειται να σταματήσουν για να πάνε στο νοσοκομείο. Πρέπει να καινοτομήσουμε λοιπόν και εμεί λόγω τη ιδιαίτερη φύση τη κρίση και τη ταχύτητα μετακίνηση των πληθυσμών. Τέλο, από τι κατευθυντήριε γραμμέ να σα διαβάσω ότι η αποτυχία μας να αντιμετωπίσουμε το περιστατικά σημαίνει μια ανθρωπιστική κρίση. Θα θετήσουμε τη βασική μα ευθύνη να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ευάλωτων πληθυσμών. Κάτι λοιπόν πρέπει να κάνουμε, να βοηθήσουμε γυναίκες και νεαρά κορίτσια για να μην αθετήσουμε την βασική μας υποχρέωση, να τις φροντίσουμε με τρόπο υπεύθυνο και ασφαλή. Η έκθεση, είναι, η έκθεση έχουμε και το ψήσιμο το οποίο εκφράζω την ικανοποίησή μου. Το θέμα είναι πάντως στην πράξη θα κάνουμε για, αυτά, για αυτούς τους ανθρώπους στο πλαίσιο της κρίσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να εσωματωθεί πιστεύω στο σχετικό ψήφισμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω απλώς ότι η έκθεση μετά από την επίσκεψή μας θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες μόλις μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, the next speaker... Ευχαριστώ, τον συμμελητής για την Παρα Σίνγκερ από την οργάνωση Asylum Aid από το Λονδίνο.

Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να έρθω σε αυτήν την ακρόαση σήμερα. Εμεί ε, έχουμε πάντα ανέκαθεν ενθαρρυνθεί ότι αυτή η Επιτροπή, η Επιτροπή των Γυναικών, ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τις γυναίκες πρόσφυγες εδώ και αρκετές δεκαετίες μάλιστα. Θα θέλαμε επίσης να καλωσορίσουμε την έκθεση της κυρίας Χάνιμπολ που συζητάμε σήμερα εδώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω σε μια συγκεκριμένη πτυχή αυτή τη έκθεση που έχει να κάνει με τι διαδικασίε ασύλου. Όταν οι γυναίκε δηλαδή που ακούσαμε τι ιστορίε του έχουν φτάσει στην Ευρώπη και έχουν καταλήξει σε μια χώρα που ζητούν άσυλο, χρειάζεται να περάσουν από μια διαδικασία ασύλου και με χαρά βλέπω ότι στην έκθεση γίνεται λόγος για διάφορες διαδικασίες και διάφορα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τις γυναίκες. Αυτό που θα κάνω λοιπόν είναι να ανατρέξω αυτές τις διαδικασίες και να εξηγήσω το, η λογική που κρύβεται πίσω από αυτές και πώς θα ωφελήσουν τις γυναίκες όταν αυτές θα έχουν πια το καθεστώς ασύλου. Καταρχήν το δικαίωμα να ζητήσουν συνομιλητή γυναίκα και διερμηνέα γυναίκα και όλοι θα καταλαβαίνετε βέβαια ότι είναι πιο εύκολο για τις γυναίκες να μιλήσουν για αυτές τις εμπειρίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σεξουαλική βία, βιασμό, οικογενειακή βία, εγχώρια, ε, ε, ενδοοικογενειακή βία, ακροτηριασμό για την οργάνων. Είναι πολύ πιο εύκολο για αυτές αν έχουν γυναίκα συνομιλητή και γυναίκα διερμηνέα. Επίσης, Έχουμε πρόσφατα δημοσίευσε μια ανέκθεση το 2012 για την ε, βία κατά των γυναικών. Συντάχθηκε από πέντε όπως συμπεριλαμβανομένες της δικής μας, ε, και εκεί συγκεντρώσαμε στοιχεία για τις γυναίκες πρόσφυγες. Στις περισσότερες χώρες ε, όντως προσφέρεται γυναίκα συνομιλητής, αλλά όχι πάντοτε διερμηνέας γυναίκα. Και επίσης οι γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να ζητήσουν γυναίκα συνομιλητή Οπότε πρέπει αυτό το δικαίωμά τους να ε, γνωστοποιηθεί περισσότερο, να πάρει περισσότερη δημοσιότητα. Η επόμενη διαδικασία για την οποία επίσης έχουμε μιλήσει αφορά την παροχή φροντίδας παιδιών στη διάρκεια των ε, συνεντεύξεων για το άσυλο. Εδώ στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, οι βελγικές αρχές ε, προσφέρουν την φροντίδα για τα παιδιά εδώ και πάνω από μια δεκαετία στη διάρκεια των ακροματικών δικασιών. Όταν δηλαδή μια γυναίκα δεν έχει να επιλέξει ανάμεσα στο να τραυματίσει το παιδί της και να, ή να μην πει ό,τι πρέπει να πει σε μια διαδικασία συνέντευξης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, επίσης ε, υπάρχει πλέον ε, τέτοιου είδους δομή για τη φροντίδα των παιδιών, αλλά στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σπάνιο. Επόμενη παρατήρηση αφορά την κατάρτιση για τους συνομιλητές και τους διερμηνείς σε σχέση με το, τη σεξουαλική βία, το τραύμα και την μνήμη και θα έρθω σε αυτό αργότερα. Έπειτα, ε, παροχή συμβουλών και παροχή πληροφοριών σε σχέση με τη διαδικασία ασύλου είναι οι διάφοροι τομείς. Τώρα, μπορεί αυτής, αυτές οι, οι εικόνες να σας εντυπωσιάζουν. Στο Ενωμένο Βασίλειο γίνεται μια εκστρατεία που ε, ονομάζεται ε, χάσμα προστασίας ε, και σχετική εκστρατεία και πολλές, ε, μια γυναίκα η οποία είναι καλλιτέχνης έχει σχεδιάσει τα λογότυπα και η εκστρατεία τρέχει εδώ και ένα χρόνο και το Υπουργείο Στερικών εργάζεται για την εγκαθίδρυση όλων αυτών των διαδικασιών που σας ανέφερα αλλά δεν επιλέξαμε αυτές τις ε, διαδικασίες τελείως τυχαία. Υπάρχει λογική πίσω από όλα αυτά και αυτό είναι ότι όλες αναφέρονται σε τρία διαφορετικά διεθνή πρωτόκολλα. Το πρώτο είναι το Διεθνές Πρωτόκολλο για την διερεύνηση και την τεκμηρίωση της σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις ε, στις σειράξεις. Και αυτό προέκυψε από την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορφής που διοργάνωσαν η Αντζελίνα Ζολή και ο Βίλιαμ Χέικ το προπέρσινο ε, καλοκαίρι στο Λονδίνο. Νομίζουμε πως είναι ηρωνικό τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πρωτόκολλο μπορούν να είναι διαθέσιμα για μια γυναίκα η οποία είναι θύμα βιασμού ως όπλο πολέμου, ας πούμε στο Κονγκό ή στη Σομαλία, ενώ δεν μπορεί να θεωρηθεί εγγυημένο για την ίδια γυναίκα εάν ε, έφτασε στην Ευρώπη και ζητά το άσυλο εδώ. Το επόμενο πρωτόκολλο είναι η οδηγία της Ένωσης για τα θύματα που άρχισε να ισχύει πριν από τρεις εβδομάδες και αν, έχει, και και έχει συνταχθεί βασικά για τις γυναίκες που είναι θύματα ε, εγκλήματος ή σεξουαλικής βίας στην Ευρώπη μπορεί να επεκταθεί για να ισχύσει και για τις γυναίκες που έπεσαν θύματα σεξουαλικής βίας σε χώρες εκτός της Ένωσης όταν αυτές φτάσουν στην Ένωση και ζητήσουν προστασία. Και έπειτα το τρίτο είναι από, το Ηνωμένο, από τα Ηνωμένα Έθνη, την Επιτροπή Γυναικών και τη σύμβαση που συνδέει τα θέματα τα προσφυγικά με τα γυναικεία θέματα. Όλα λοιπόν τα μέτρα που ανέφερα και περιλαμβάνονται στην έκθεση της κυρίας Χάνιμπολ, στη σελίδα 9, αν τα ψάχνετε, περιλαμβάνονται σε αυτά τα πρωτόκολλα. Υπάρχει λοιπόν διεθνή νομική βάση από τα διεθνή αυτά πρωτόκολλα απορρέει από τα διεθνή αυτά πρωτόκολλα, αλλά λείπουν από τα συστήματα ασύλου της Ευρώπης. Και για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά τα μέτρα. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση που δώσαμε που δείχνει ότι η αξιοπιστία είναι στον πυρήνα της άρνησης του ασύλου στις περισσότερες γυναίκες. Δηλαδή δεν τους χορηγείται το άσυλο επειδή δεν τους πιστεύουν. Και αυτό φυσικά επαναφέρει το θέμα της σημασίας της αξιοπιστίας που το αναφέρετε και εσείς στο έγγραφό σας. Το θέμα της αξιοπιστίας φυσικά προκύπτει και στην Ευρωπαϊκή Έκθεση που εσείς δημοσιεύετε, που εμείς μάλλον δημοσιεύσαμε και αναφέρεται και στην έκθεση της UNHCR που λέει πέρα από τις αποδείξεις και μιλά για τη διαδικασία τη αξιοπιστίας και επίσης αναφέρεται και στις δικές μας έρευνες που κάναμε ε, όπου διαπιστώσαμε ότι όταν στις γυναίκες δεν δίνονταν άσυλο ήταν, οφειλόταν πάντοτε σε δυσπιστία και επειδή συχνά ανατρεπόταν μετά από έφεση γιατί ακριβώς ο ειδικό δικαστής για τη μετανάστευση τους πίστευε. Είχαν δηλαδή διαφορετική αξιολόγηση αξιοπιστίας στην φάση της έφεσης διαπιστώσαμε ότι αν είσαι γυναίκα είναι πιο πιθανό να ανατραπεί η απόφαση στο εφετείο α, α, α, περισσότερο πιθανό μάλλον να ανατραπεί η απόφαση στο εφετείο αν είσαι γυναίκα από ότι αν είσαι άνδρας. Υπάρχει ένα βιβλίο στο, το οποίο λέγεται «Το φίλο στην ε, νομοθεσία περί προσφύγων» και βρίσκεται και σε ένα φίλο που φτιάξαμε εμείς στο Asylum Aid το οποίο θα κυκλοφορήσει από το γραφείο της κυρίας Hannibal. Η ανάλυση μας είναι λοιπόν ότι υπάρχουν τρεις αλληλένδετοι, μάλλον σχετιζόμενοι παράγοντες που οδηγούν στην ε, δυσκολία της αξιοπιστίας ε, της γυναίκας. Δηλαδή το, οι αποδείξεις, οι αποδείξεις ερμηνεύονται εξαιρετικά αυστηρά στα αιτήματα ε, ασύλου της, ε, των γυναικών και αυτό εν μέρει επειδή είναι πιο δύσκολο για τις γυναίκες να έχουν τεκμηριωμένες αποδείξεις για να αποδείξουν ε, το αίτημα ασύλου. Αν σκεφτείτε έναν άνδρα πολιτικό ακτιβιστή μπορεί να έχει κάρτα μέλους ή μπορεί να έχει μια φωτογραφία ότι συμμετέχει σε διαδηλώσεις. Αλλά οι γυναίκες πολιτικές ακτιβίστριες πολύ συχνά συμμετέχουν με διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί ας πούμε να προσφέρουν τρόφι και ε, κατάλημα στους άνδρες και δεν έχουν τεκμηριωμένες αποδείξεις γι' αυτό. Και για τις γυναίκες που διώκονται λόγω φύλου, ε, πίστη είναι δύσκολο να έχουν αποδείξει. Δεν έχει κανεί πιστοποιητικό επειδή το χτυπάνε σπίτι του και επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν αποδείξεις, οι γυναίκες ε, βασίζονται στη προφορική μαρτύρια. Και επειδή αυτό το θέμα έχει να κάνει με το τραύμα που ανέφερα πριν και που επηρεάζει τη μνήμη τους και την τροπή που νιώθουν, καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο να διηγηθούν τι τους έχει συμβεί. Δίνουν λοιπόν συνήθως μαρτυρία η οποία δεν είναι συνεπής, περιέχει κενά, και βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου αυτοί οι τρεις παράγοντες ε, συσχετίζονται μεταξύ τους και δημιουργούν μια πραγματική δυσκολία για τις γυναίκες στόν να έχουν θετική αξιολόγηση και ακριβή αξιολόγηση αξιοπιστίας. Τα μέτρα για τα οποία λοιπόν μίλησα θα βοηθήσουν στο να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια θετική ή ακριβή ε, ε, μελέτη αξιοπιστίας, μάλλον αξιολόγηση αξιοπιστίας και θα δείτε ότι στη δήλωση, αλλά θα πρέπει να είναι κατά τη γνώμη και στο ψήφισμα, στα ψηφίσματά σας να λέει λοιπόν ότι καταρχήν οι διαδικασίες θα βοηθήσουν στις γυναίκες να ξεπεράσουν την έλλειψη ε, ε, αποδείξεων, αποδεικτικών στοιχείων και θα τις βοηθήσουν να δείξουν ότι η μαρτυρία τους είναι συνεπής και ολοκληρωμένη. Εάν λοιπόν ληφθούν αυτά τα μέτρα θα σήμαινε ότι θα είμαστε σε καλύτερη θέση για να εναρμονίσουμε τις προδιαγραφές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως ξέρετε, πολύ ε, διαφέρουν αυτή τη στιγμή οι προδιαγραφές θα έχουμε ε, κοινέ γραμμές, όπως προτείνει και η κυρία ε, Χάνιμπολ, και θα είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να έχουν ε, ακριβείς αξιολογήσεις αξιοπιστία για να μπορούν να έχουν δίκαιες αποφάσεις ασύλου και μάλιστα με την πρώτη φορά κατευθείαν. Η σωστή λοιπόν αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική για τις γυναίκες που έρχονται στην Ευρώπη για να αναζητήσουν προστασία, ε, κατά των ε, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες τους. Ευχαριστώ. Εγώ αναλαμβάνω τώρα τα ενία της ε, διευθύνσεως της συζήτησης, λέει η κυρία Χάνι και η επομένη ομιλήτρια θα είναι η κυρία Σιέσιο από το Μάλμο της Σουηδίας και ε, θα εξηγήσει ε, μια προσπάθεια που κάνουν εκεί για να βοηθήσουν γυναίκες πρόσφυγες. Thank Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, διότι όλο το εγχείρημα που ξεκίνησε με χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και που λέγεται Γιάννα Τράπαν και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη μέσω ε, κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για μια ε, συνεργασία γυναικών, για ένα συνεταιρισμό γυναικών ε, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με χαρακτηριστικά την συμμετοχή και το empowerment, την ε, ενδυνάμωση των εισαγωγικών. Γιατί εκεί πιο σημαντικά πράγματα αυτά από την αποκόμιση κέρδους. Η άλλα Τράπαν έχει κοστίσει 8 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες το κράτος, ε, για την περιφέρεια και για την ε, ε, τοπική κοινότητα εδώ και τέσσερα χρόνια. Ο στόχος είναι οι γυναίκες που συμμετέχουν να αισθάνονται καλά και τα παιδιά και τα λοιπά και να μπορούν να βγάλουν και κάποια χρήματα. Είπα ότι δεν κυνηγάμε το κέρδος, αλλά υπάρχει χώρος για συμμετοχή, για έργο στο επίπεδο της κοινότητας και για δημοκρατία. Η ομάδα στόχος της Γιάλα Τράπαν είναι γυναίκες που διαμένουν στο Ρούσονγκορ, στο Μάλμε, με περιοχή με υψηλό ποσοστό μεταναστριών και υψηλό ποσοστό ανεργίας. Ε, οι γυναίκες αυτές έχουν έλλειψη προσόντων και εκπαίδευση που να είναι κατάλληλα και για τη Σουηδία αλλά και από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Δεν γνωρίζουν καλά τη σουηδική γλώσσα και είναι εντελώ εκτός της αγορά εργασίας. Έχουν ζήσει ορισμένε από αυτές πολλά χρόνια στην Σουηδία και έχουν ε, πολύ συχνά ε, άδειε ασθένεια. Συνεργαζόμαστε μαζί τους και για την εκπαίδευση, συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες και συνεργασία και μέσα σε μικρές επιχειρήσεις συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη ή ε, στην τοπική κοινωνία, μαθήματα σουηδικής γλώσσας και ε, διάφορες, διάφορα καθήκοντα που αναλαμβάνουν. Τώρα, ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα. Μετά από ένα χρόνο βλέπουμε ότι όταν οι γυναίκες έχουν έρθει από την αρχή με ε, χαμηλή αυτοπεποίθηση, και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και έχουν μια υπερηφάνεια επειδή έχουν μια απασχόληση και ανακτούν μια αξιοπρέπεια όλο τον καιρό που έχουν ζήσει στη Σουηδία και εξαρτώνται απολύτως από επιδόματα ενώ τώρα αρχίζουν και ε, αποκτούν χρήματα δικά τους από μακρόχρονες ε, ε, περιόδους ασθενείας, αδειές ασθενείας δηλαδή, τώρα είναι, πολύ πιο σπάνιες αυτές χρησιμοποιούν πολύ λιγότερα φάρμακα. Ενώ έχουν ξεκινήσει από σπάνιες κοινωνικές επαφές, τώρα αυτές έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Ήταν άρρωστες, τώρα είναι υγιείς. Και κάτω εκεί στην φωτογραφία αριστερά βλέπετε τον Μοχάμετ Γιούνας, ε, βραβευμένο με βραφείο Νομπέλ, που ήρθε και μας επισκέφθηκε. Εργάζεται πολύ και ε, γι' αυτό το αναφέρω άλλωστε για ε, μικρές κοινωνικές, υπέρ μικρών κοινωνικών επιχειρήσεων. Άλλη θετική έκβαση είναι ότι οι γυναίκες αυτές από το να είναι εντελώ ανώνυμες να αρχίσουν να τις βλέπουν πλέον στην κοινωνική ζωή, συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. Δεν ψήφιζαν ποτέ, τώρα όλες πηγαίνουν και ψηφίζουν. Και ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι έχοντας ξεκινήσει από μια πολύ αδύναμη θέση στις πατρίδες τους, τώρα γίνονται πραγματικά παραδείγματα για τα παιδιά τους. Ξέφυγαν από την μοναξιά και τη μοναχικότητα και έχουν ενταχθεί σε κοινωνικό έργο ε, από εκεί που δεν είχαν απολύτως καμία ισχύ τώρα ε, έχουν ενδυναμωθεί. Αυτός είναι και ο στόχος του συνεταιρισμού μας, άλλωστε ε, η δημοκρατική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Μέσα στη αλλά και πέρα από τα όρια της κοινότητας ε, Ουσενγκότ, έχουμε φτάσει και στην Ισταμπούλ, όλοι μαζί, για πρώτη φορά και χωρίς γυναίκες και παιδιά. Ωραίο ταξίδι αυτό. Και βέβαια, από εκεί που αισθάνονταν να μην έχουν καμιά αξία, τώρα αισθάνονται ότι οι άλλοι άνθρωποι τις έχουν ανάγκη και ότι μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Η ε, ε, εμπορική κράτη της Γιάλα Τσάπαν Φαίνεται πως υπάρχει κάποιος θόρυβος πίσω. Ε, προσφέρουμε υπηρεσίες ε, καφενείων, ε, catering, φτιάχνουμε μαρμελάδες, προσφέρουμε υπηρεσίες καθαρισμού. Με συγχωρείτε εδώ κάτι έγινε με τη διαφάνεια. Επίσης έχουμε ένα στούντιο. Κάνουμε και, μάλλον δεχόμαστε επισκέψεις μελετητών κάθε μέρα, κάνουμε και ξεναγήσεις. Έχουμε γράψει δύο βιβλία. Το ένα λέγεται The Road to Yala. Εκεί περιγράφουν τη ζωή τους οι ίδιες οι γυναίκες, πώς έφτασαν μέχρι εκεί ως πρόσφυγες, μέχρι σε εμάς δηλαδή. Και το άλλο λέγεται Yala Trapan, So We Did It. Έτσι τα καταφέραμε. Και είναι ένα βιβλίο που θα το χρησιμοποιήσουν όλοι και να διδαχθούν κάτι από αυτό η δομή μας έχει ως εξής, όπως την βλέπετε. Έχουμε και γραφεία με ε, υπαλλήλου. Ήταν ε, αρχικά 8. Έξι από αυτούς ε, είχαν μόνο 25% του χρόνου απασχόλησης. Και τώρα μετά από 4 χρόνια έχουμε φτάσει στους 29 και οι περισσότεροι, οι περισσότερες από τις εργαζόμενες αυτές έχουν η πλήρη απασχόληση 75%. Έχουμε και εκπαιδευομένους με τις ίδιες γυναίκες, με τις ίδιες τις γυναίκες του Γιάννα Τράπαν. Έχουμε και συμφωνίες με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα με τον καλύτερο τρόπο τις νέες εκπαιδευόμενες γιατί έχουν περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία οι ίδιες οι γυναίκες μας. Στο στούντιο ε, ασχολούμεθα ιδίω με την ανακύκλωση. Έχουμε και μια συμφωνία με μια μεγάλη επιχείρηση για προσφορά υπηρεσιών, μόνο η Σουηδία. Μετά από αυτά τα πέντε χρόνια τώρα μετακινήσαμε το στούντιό μας για τρίτη φορά διότι γίνεται όλο και δηλαδή γίνεται ξανά και ξανά μας φαίνεται μικρό και ε, στην κουζίνα έχουμε όπως είπα catering, φτιάχνουμε μαρμελάδες και βέβαια με ε, γεύσεις της Μέσης Ανατολής και βέβαια κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις. Οι υπηρεσίες καθαρισμού και ε, συναντήσεων συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείε και, άλλους, ε, και άλλες οργανώσεις, κυρίως για τον καθαρισμό γραφείων. Έχουμε 10 πελάτες. Όλα όσα σας εξηγώ τώρα τα έχουμε κάνει όλες μαζί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή οι πρόσφυγες μαζί με ε, εμάς. Προσπαθούμε επίσης να βελτιωνόμαστε, να αναπτυσσόμεθα δηλαδή διαρκώς Έχουμε και μια, οργάνωση, μια συνεργασία μάλλον με την κοινότητα Μάλμε, Γιάλας Road to Work, τη λέμε στα αγγλικά. 40 γυναίκες τον χρόνο εκπαιδεύονται σε θέματα ε, εργασίας και επίσης σε θέματα ε, μαγειρικής κλπ. Και έχουμε και τους Γιάλας Ambassadors, τους πρέσβεις της Γιάλα και η συμμετοχή μας ε, στην πρόθεση κοινωνικών επιχειρήσεων μαζί με την ΕΒΕΦ και το κοινωνικό ταμείο της Ινσκιώνα που είναι άλλη πόλη στο νότο της ε, Σουηδίας θέλουμε να ξεκινήσουμε μια άλλη οργάνωση ένα άλλο γραφείο δηλαδή το βιβλίο που ανέφερα πριν, Yala So We Did It, πολίτες σε 60 άλλες κοινότητες που όλες αντιμετωπίζουμε την ίδια πρόκληση. Ε, ε, ε, και αυτό εξαρτάται από, το, από ποια χώρα προερχόμαστε. Τέλος, νομίζω ότι επιτύχαμε διότι στοχεύσαμε στα κοινά στοιχεία όλων αυτών των γυναικών και παρά τις διαφορές τους οικονομικές, κοινωνικές, ε, εθνικές και άλλες και βασιστήκαμε επίσης στους ίδιους τους, τους των γυναικών αυτών. Τους δίνουμε τα μέσα και την ευκαιρία να αλλάξουν και να προσαρμοστούν. Σας ευχαριστώ. Thank you. I'm sure you'll... Σας ευχαριστώ. Είμαι βεβαία ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ήταν ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις και προσφέρουν νέα στοιχεία στην συζήτηση. Πριν δώσω το λόγο σε άλλα μέλη, θα δώσω πρώτα στην κυρία Κιένγκε, που είναι η συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής ε, Θεμελιωδών Ελευθεριών. Κυρία Κιένγκε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την δημόσια κρόση. Για μένα είναι χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σας σε αυτή την στιγμή και να ακούσω τους εμπειρογνώμονε και όλες τις εισηγήσει που παρουσιάστηκαν. Δεν θα σας πω μόνο ε, προσωπικές απόψεις, αλλά θα προσπαθήσω να εντάξω τις δικές σας ε, συμβολές ε, στην ε, έκθεση πρωτοβουλίας για την οποία είμαι συνεισηγήτρια, της οποίας τίτλος είναι «Η κατάσταση στη Μεσόγειο» και ανάγκη μιας σερικής ολιστικής προσέγγισης στο μεταναστευτικό φαινόμενο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ήταν για μένα να είμαι σήμερα εδώ, να σας ακούσω και να μπορέσω να χρησιμοποιήσω τις συμβολές σας στην εργασία αυτή. Το θέμα που αντιμετωπίζετε σήμερα μου είναι ιδιαίτερα αγαπητό και πάντοτε αισθανόμουν προσωπική δέσμευση και προσήλωση σε αυτό το θέμα. Ε, από το παρελθόν που έχω παρέμβει για το θέμα των γυναικών και ήμουν η πρώτη, μία από τις πρώτες που στήριξαν το πρωτόκολλο του Μαπούτο που είναι ο χάρτης για την αξιοπρέπεια και την και τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι θεμελιώδης για τις αφρικανικές, αφρικανές γυναίκες. Αυτό το πρωτόκολλο, αυτός ο χάρτης έχει μεγάλη σημασία γιατί έχει προωθηθεί από τις ίδιες τις γυναίκες της Αφρικανικής Υπήρου που κατέστησαν κατανοητές τις ανάγκες τους και κατάφεραν επίσης να το, να το τοποθετήσουν εντός ενός εγγράφου, ενός δοκουμέντου της Αφρικανικής Ένωσης. Δυστυχώς αυτό το έγγραφο έχει υπογραφεί από 15 χώρες, έχει κυρωθεί μόνο από 28, όπως καταλαβαίνετε μένει πολλή δουλειά ακόμα. Το σχέδιο τώρα έκθεση τη συναδέλφου Μέρι Χόνιμπολ περιγράφει ε, με μεγάλη ακρίβεια την κατάσταση στην οποία βρίσκονται εκατοντάδε χιλιάδες γυναίκε ε, και κορίτσια και που αναζητούν ε, διεθνή προστασία στι χώρες μέλη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εργαστούμε. Οι γυναίκες που ζητούν άσυλο χρειάζονται ειδική προστασία και διαφορετική από αυτή των ανδρών. Αυτό, πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Σε κάθε έκθεση και σε κάθε τομέα που αγγίζουμε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότερες γυναίκες που είναι φυγάδες δεν θα καταφέρνουν να ζητήσουν άσυλο στο εξωτερικό και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί ο δρόμος τους πολύ νωρίτερα σταματά διότι ορισμένες γυναίκες υπόκειται σε βία ακόμα πριν μπορέσουν και προλάβουν να βάλουν το πόδι στη χώρα προορισμού τους. Ωστόσο, ούτε για αυτές που φτάνουν, ε, που τα καταφέρνουν, το άσυλο είναι πάντα συνώνυμο της σωτηρίας. Η σεξουαλική βία, η βία που οφείλεται στο φύλλο δεν γίνεται μόνο στις χώρες προέλευσης ή στις χώρες διέλευσης, συνεχίζεται και στις χώρες υποδοχής και το δράμα που ζουν οι γυναίκες ε, από τη στιγμή που αποφασίζουν να φύγουν από τις χώρες τους, σε όλη την πορεία και συνεχίζεται και στη χώρα υποδοχής. Μέχρι στιγμή τα συστήματα ασύλου σε μεγάλο τμήμα έχουν αξιολογηθεί μόνο από την ανδρική οπτική. Και εγώ πιστεύω πως πρέπει να ξεφύγουμε από αυτήν την ε, στάση. ή και, η ώρα να αλλάξουμε δραστικά πορεία, Ρώτα. Η εφαρμογή των πολιτικών μας σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το θέμα του φύλου. Συχνά έχουν υπάρξει διδασκολίες για τις γυναίκες να γίνουν κατανοητές, να επιμείνουν για τις δικές τους ανάγκες και πολλές φορές ταπεινώνονται κιόλα. Ίσως μια γυναίκα που έχει υποστεί βία τη ζητούν να δώσει αποδείξεις είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια γυναίκα που, όλη, που να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ταπείνωσης. Χρειάζεται πολλές φορές και ψυχική βοήθεια, ψυχολογική βοήθεια και κυρίως να καταργηθεί κάθε είδος συντήρησης ε, γυναικών ε, εγγύων που έχουν υποστεί τραύματα ή ε, βία οποιοδήποτε είδους να, θα πρέπει στη διάρκεια της διαδικασίας να τους εγγυηθούμε ε, γυναικεία βοήθεια και κυρίως ε, στην κοινωνική ένταξη και στην ε, ένταξη την κοινωνική, να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη παιδεία και στην αγορά εργασία και οι δικέ σα συμβουλέ ήταν πολύ σημαντικέ γιατί καταστούν κατανοητή τη σημασία της ένταξη και τη πρόσβαση στην εργασία. Θα ήθελα ωστόσο κάτι να πω και να συγκεκριμενοποιήσω κάπως αυτό που λέει και η συνάδελφος Μέρη στην ε, έκθεσή της. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, οδοί πρόσβασης ασφαλής και νόμιμες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια αρχή που έχουμε εντάξει ξεκάθαρα και στο δική μας ε, έκθεση πρωτοβουλίας. Επιτρέψτε μου μια τελευταία μνήμα στην ε, κατάσταση των γυναικών και στις δίκες των γυναικών, ε, των γυναικών. Μόλις επέστρεψα από την Κουρκίνα Φάσο, όπου επικεφαλής ε, της αποστολής παρατήρησης των εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήμουν εγώ και παρακολούθησα την έκφαση των εκλογών για λογαριασμό της Ένωσης. Μπόρεσα να διαπιστώσω από πρώτο χέρι την βούληση και τη δέσμευση των γυναικών, τη συμβολή τους και τη συμμετοχή τους στο εσωτερικό της κοινωνίας των πολιτών. Δυστυχώς αυτό που λείπει ακόμα είναι η πλήρη του συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Το γεγονός ότι ακόμα αποκλείονται από τις δυνατότητες και τους αρνούνται τα υψηλές θέσεις στην λήψη αποφάσεων. Στις 14 υποψήφιους μόνο δύο ήταν γυναίκες και με ελάχιστε δυνατότητε εκλογή. Αυτή η κατάσταση δεν είναι πια αποδεκτή. Εγώ μίλησα με διάφορε οργανώσει και ανάμεσα στι δικέ μα αναλυτέ τη ομάδα που είχαμε δηλαδή μαζί, υπήρχε και μια αναλύτρια που ασχολείται με θέματα φύλου και μα έδωσε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε και σε αυτό το θέμα. Θεωρώ πως η χειραφέτηση των γυναικών περνά και από την πλήρη του συμμετοχή στην δημοκρατική ζωή και στην θεσμική ζωή της χώρας τους. Νομίζω πως με αυτή τη σύντομη παρέμβαση και ευχαριστώντας ακόμα μια φορά τη συνάδελφό μου και κυρίως αναγνωρίζοντας τη σημασία του σχεδίου έκθεσης της, θα ήθελα άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους και ελπίζω ότι θα μπορέσω να διαβιβάσω και τις δικές σας ε, παρεμβάσεις στη δική μου επιτροπή. Oh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, εισηγήση των σκιωδών. Παρακαλώ κύριε Κόατσα Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την Μπάρμπαρα Ματέρα, η οποία δυστυχώ δεν μπορεί να παρευρεθεί που είναι η σκιώδη, αλλά πριν ξεκινήσω να πω προς όλες σας ότι ήταν πραγματικά πολύ εμπρευστικές οι ομιλίε. σας. Θα τα μεταφέρω φυσικά στην Βάρβαρα αλλά και στο ΕΛΚ. Όλα αυτά τα σημαντικά που μα είπατε. Θα προσπαθήσω και εγώ να συνεισφέρω στην εξαιρετική, ε, στο εξαιρετικό έργο της υπότης και των ΜΚΟ. Τα γνωρίζουμε αυτά στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ και την Χριστίνα, η οποία είναι από τη Σουηδία. Είχα πάει στο Μάλμα. Η Ροζενκορ στιγματίστηκε ως ε, μια από τις δυσκολότερες περιοχές για επανεσωμάτωση ε, χαρακτηριστική ως γκέτο και εσείς από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο ήταν τα πράγματα να χειριστείτε περιοχές περιθωριοποιημένες. Μερικές φορές οι κοινωνίες μας πετυχαίνουν χάρη στη δύναμη των γυναικών να γίνουν υποδείγματα ενσωμάτωσης πραγματικά εντυπωσιάστηκα όταν επισκέφθηκα την περιοχή. Ελπίζω ότι το προηγούμενο αυτό θα μα βοηθήσει και εμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγγνώμη για την παρέκβαση, αλλά ήθελα να πω δύο πράγματα τα οποία θεωρούσα σημαντικά. Λοιπόν, ένα ευχαριστώ καταρχά στην κυρία Χάνιμπολ για το εξαιρετικό έργο τη, την εξαιρετική έκθεση. Ναι, η ενσωμάτωση τη διάσταση του φίλου στι πολιτικέ μα είναι πολύ σημαντικό. Και δι, ε, το πρόβλημα των μεταναστών και προσφύγων. Πάρα πολύ σημαντικό για όλου του λόγου που μόλι αναφέραμε. Πολλέ φορέ, τι περισσότερε μάλλον φορέ, η βία προέρχεται από άνδρε και τα θύματα είναι γυναίκε και παιδιά. Για να μην μιλήσω για την βία, για τον ακροτηριασμό των γενικών γενετικών οργάνων κλπ. Υπάρχει το θέμα του τράφικινγκ, του εμπορίου ανθρώπων, που πλήττει κυρίω τι γυναίκε, Είναι προφανέ το πρόβλημα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Πρόκειται για τράφικινγκ με σκοπό την πορνεία και την σεξουαλική εκμετάλλευση. Πρέπει να καλέσουμε όλα τα κρατημέλη να ακυρώσουν τι σχετικέ συμβάσει για την βία κατά των γυναικών. Και να υποστηρίξουμε βεβαίω την ανάγκη συλλογή στοιχείων σε αρτήση του φίλου τώρα με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Η Μπάρμπαρα πιστεύει επίσης ότι πολλά θέματα παρ' όλα αυτά είναι το μάλλον της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, είναι θέματα σύλλου ή των κρατών μελών βάσει επικουρικότητας. Στην παράγραφο 7 που αναφέρεται πολλές από εσάς, σε λεπτό κάπου εδώ έχω γράψει κάτι για την παραγραφή 7. ο κατάλογος των ασφαλών χωρών. Δεν ακυρώνει το γεγονός ότι το πακέτο ή το άσυλο αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο, αφορά το πρόσωπο. Δηλαδή, ακόμη και αν προέρχεσαι από ασφαλή χώρα, μπορεί όντως να έχει δικαίωμα παροχής ασύλου βάσει της ε, συγκεκριμένη αξιολόγηση. Και εκεί δεν ισχύει η αρχή της επαναπρόθεσης ούτε έχει νόημα να χωρίσουμε τι χώρε σε των κινδύνων που αντιμετωπίζουν άντρε και γυναίκε. Και είναι και δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Επίση, πιστεύει η Μπάρμπαρα ότι ήδη στη δέσμη για το άσυλο υπάρχουν διατάξει για τι ευάλωτε ομάδε για θύματα βασανιστήριων, ακροτηρισμού γεννητικών οργάνων, βιασμού και άλλων συναφών πράξεων που είναι σε αρτήση του φύλου στη για το άσυλο. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να λυθούν υπόψη. Στην παράγραφο 10 υπογραμμίζει ότι έχει σημασία, όπως άλλωστε το είπατε και εσεί, την σημασία οι συνεντεύξεις να διεξάγονται από γυναίκες διερμηνεί και ακόμη περισσότερο από εκπαιδευμένου ανθρώπους. Παράγραφο 9. Βαρβαρά είναι υπέρ της διαφάνειας και τη συλλογή στοιχείων. Πιστεύει όμω ότι θα είναι πολύ δύσκολο αυτό, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, τα κράτη-μέλη δηλαδή, να τηρούν στατιστικέ ε, για τι θετικέ περιπτώσει, θετικέ απαντήσει για γυναίκες. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να συλλογούν οποιαδήποτε στοιχεία. καταστάσει κράτηση. Ξέρετε, στο κείμενο γράφεται detention facility, εγκατάσταση κράτηση Μήπως υπάρχει εδώ μια σύγχυση, άλλο εγκατάσταση υποδοχής, άλλο εγκατάσταση κράτησης, άλλο εγκατάσταση φιλοξενίας, όλα αυτά να γράψουμε καλύτερα κέντρα υποδοχής. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται. Παράγραφος 14, πρόσβαση σε δημοσιογράφους, το λέει και η αυτό, μετά η διάρκεια των, της κράτησης για τους σκοπούς της εξαίρεσης της αιτησίας ασύλου, επανένωση οικογενειών, η Επιτροπή θα... Κοιτάξτε, δεν υπάρχει λόγο να συζητήσει όλο το θέμα του ασύλου ξανά από την αρχή. Δεν είναι δική μα αρμοδιότητα. Η Μπάρμπαρα λέει να επικεντρωθούμε στα θέματα του φίλου. Και αν. Ε, γιατί θέλω να μιλήσω και εξ ονόματό μου, να τα πω τώρα ή να τα πω μετά. Τι, τι θέλετε. Όχι, όχι, σε λίγο. Τώρα μιλούν ουσιαστικά οι σκιώδει. Πολύ ωραία. Αυτά εκ μέρου τη σκιώδου τη κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπορκ από την Γκουα, επόμενη σκιώδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τι εμπειρογνώμονε, τι προσκεκλημένε. Έμαθα πολλά από αυτέ εδώ, ω εκπρόσωπο της Γκουε. Και να ευχαριστώ στην ε, κυρία Μπόλ, Εξαιρετικό κείμενο. Η εφητερία για μας είναι ότι το πακέτο ασύλου υφίσταται, δεν είναι αρκετά χρήσιμο όμως για τις γυναίκες. Γι' αυτό και εμείς διατυπώνουμε συστάσεις για το πώς πρέπει να διατυπωθεί για να έχει και κάποιο αποτέλεσμα για τις γυναίκες. Θα μπορούσε κάποιο να πει, να ισχυριστεί ότι δεν αποδίδει καθόλου το πακέτο για τους πρόσφυγες ούτως ή άλλως, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, εγώ από τη Σουηδία και θα συνεχίσω στα σουηδικά. Παρακαλώ, φορέστε τα ακουστικά σας. Λοιπόν, όπως είπε και η Σίτρια, έχει πολύ μεγάλη σημασία όλες οι γυναίκες να έχουν δικαίωμα προστασίας. Σήμερα δεν υπάρχει ασφαλής δίωδος, ασφαλή διάδρομος για τις γυναίκες όταν, για τις γυναίκες που θέλουν να μπουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να στραφούμε και να κάνουμε κάτι για τις γυναίκες οι οποίες είναι στο δρόμο στην κυριολεξία και που υποβάλλουν αίτηση για άσυλο. Οι προγνώμονες μίλησαν για τους δρόμους των προσφύγων. Πρέπει να σας πω ότι με την προσωπία μας πήγα στα Δυτικά Βαλκάνια και συναντήσαμε όπως άλλωστε και πολλοί από εσά. αυτούς τους ανθρώπους. Είναι φανερό ότι χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η σεξουαλική βία. Όπως το είπατε, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν τρομακτικό άγχος και πίεση. Οι γυναίκες γεννούν στο δρόμο, στη κυριολεξία. Και βεβαίω υπάρχει και βία σε αυτούς τους δρόμους. Σεξουαλική βία. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τη βία σήμερα. Όσον αφορά τώρα τις συγκεκριμένε ανάγκες των γυναικών στα κέντρα υποδοχής, προφανώς πρέπει να λυθούν υπόψη οι ανάγκες αυτές. Πρέπει επίσης οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων να διεκπαιρώνονται έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των γυναικών. Μίλησε επίσης για εμπόριο ανθρώπων, για τράφικινγκ. Οι γυναίκες είναι πάρα πολύ συχνά θύματα του τράφικινγκ και πολλές φορές μάλιστα πρέπει να σας πω ότι όχι μόνο υφίστανται την βία, όχι μόνο εξωθούνται στην πορνεία, αλλά μετά στέλνονται και πίσω στη χώρα τους, αφού υποστούν όλα αυτά τα δεινά. Δεν χρειάζεται και εδώ να κάνει κάτι η Ευρώπη. Κύριε Χάνιμπολ, λέει κάτι που με βρίσκει σύμφωνη. Να μπορούμε να το πετύχουμε με κάποιες τροπολογίες εδώ και εκεί. Τώρα όσον αφορά την ενσωμάτωση. Μου κίνησε το ενδιαφέρον. Μιλήσατε για την Ένωση για Λατραπάν. Τα συστήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα εννοείται, αλλά το παράδειγμα αυτό από τη Σουηδία είναι εξαιρετικό. Διότι μας αποδείξατε ότι κάποιος πραγματικά μπορεί να κάνει πολλά όταν προσφέρεται αφιλοκερδός, όταν συνεργάζεται, όταν η προσπάθεια είναι ομαδική, συλλογική και όταν όλοι συμμετέχουν σε όλη την διαδικασία. Χάρη τα όσα μας είπαν οι εμπειρογνώμονες, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια εξαιρετική έκθεση. Κύριε Συγητρία, είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε. Πιστεύω ότι την διάσταση του φίλου ακριβώς πρέπει να την τονίσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. από τους πρασίνους, είναι ο επόμενος ομιλητής. ευχαριστώ πολύ κυρία Χονιμπόλ για την εργασία σας, για την έκθεσή σας, αλλά και για την ευκαιρία που μας δώσατε απόψε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θέλω να ε, ε, πρέπει σήμερα να αντικαταστήσω τη ε, Ορτασόν και ο οποίος μόλις έγινε πατέρας και άρα συνειδητοποιεί πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσεις την ζωή ενός ευρωβουλευτή με τη ζωή ενός πατέρα. Ε, έχω εδώ όμως τις σημειώσεις του. Θα πρέπει να έχουμε επίση ε, στο υπόψη μας ότι μιλώντα, μιλάμε για το κοινό σύστημα ασύλου, το οποίο όμως δεν εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη έχει ανυψώσει τύχη φραγμούς και έχει σταματήσει τον κόσμο που θέλει να έρθει να ζητήσει αυτό το άσυλο και μάλιστα ε, τους υποχρεώνουμε, όπως είπε και η συνάδελφος, να ακολουθήσουν παράνομους δρόμους που τους ε, κάνουν να πέφτουν ε, εντό εισαγωγικών στα δίχτυα των διακινητών, των ανθρώπων που μετατρέπουν τον άνθρωπο που αναζητεί άσυλο και καταφύγιο σε παράνομο άνθρωπο. Αν και κανείς άνθρωπος δεν είναι παράνομος, πάντως κάνει κάτι παράνομο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση, διότι δεν θεσπίζει αυτά τα νόμιμα, τους νόμιμους, νόμους διάβλους ένταξης, για να μπορέσουμε να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Και επίσης ακόμα ένας αντίκτυπος είναι ότι δυστυχώς για τον Ευρωπαίο ο πρόσφυγας, ο άνθρωπος που ζητά άσυλο, θεωρείται ένας παράνομος άνθρωπος και άρα δεν τον κάνουμε παρέα, δεν τον υποδεχόμαστε, τον βλέπουμε με στραβό μάτι και άρα αυξάνεται το μίσος και η απόρρεψη απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που στην ουσία προσπαθούν να σωθούν που είναι ε, να σώσουν την ίδια τους τη ζωή, πράγμα που είναι αναφέροντο δικαίωμα για όλους μας. Αυτό το σχέδιο έκθεσης τώρα είναι πολύ αξιόλογο και σαφές και νομίζω ότι τα είδαμε σήμερα εδώ, ε, τα ακούσαμε και από τις τέσσερις εμπειρογνώμονες και θα μπορέσουμε να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο με τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας έδωσαν. Είναι ένα ε, σχέδιο για την έλλειψη στοιχείων που έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί πολλές φορές δεν καταγγέλλεται αυτή η βία που ασκείται στις γυναίκες που προσπαθούν να φτάσουν εδώ και ζητώντας ε, καταφύγιο και άσυλο. Επίσης στην έκθεσή σας σωστά μιλάτε για την έλλειψη κατάρτισης για τους ανθρώπους που θα έπρεπε να τις υποδεχτούν τόσο στα σύνορα όσο και στα κέντρα υποδοχής. Εδώ επίσης αναφέρθηκε το θέμα του καταλόγου με των ασφαλών χωρών. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή επιστρέφει σε χώρες που δεν είναι καθόλου σίγουρες ανθρώπους που προσπαθούν να ζητήσουν άσυλο ή καταφύγιο. Άρα λοιπόν πολλά, πολλούς μάλιστα πρόσφυγες δεν τους ακούμε καν. Να σας πω ότι γίνεται στη Θεούτα και στη Μελίγια, στην Ισπανία. Ε, πολλές φορές ε, επιστρέφονται άνθρωποι εν θερμό. Επιστρέφονται στο Μαρόκο αυτοί οι άνθρωποι, όπου όπως ξέρουμε είναι ένα κράτος, ε, το Μαρόκο, που δεν αναγνωρίζει την ε, σεξουαλική βία, ούτε την βία λόγω φύλου. Η βία μέσα στο γάμο δεν θεωρείται εγκλημά, δεν θεωρείται τίποτα. Η Ευρώπη δηλαδή επιστρέφει σε αυτή τη χώρα ανθρώπους χωρίς καν να ρωτοζωτήσει το όνομά τους. τους ε, στέλνουμε πίσω τελείως ανυπεράσπιστους. Δεν μπορούμε λοιπόν, είπατε κυρία Χόνιμπολ, κανέναν ε, άνθρωπο που ζητάει άσυλο να τον επιστρέψουμε σε μια χώρα όπου δεν αναγνωρίζεται σαφώς ε, η ισότητα των γυναικών και μάλιστα που δεν υπάρχει νομοθεσία κατά της βίας ε, σεξουαλικού τύπου υποφίλεται στο φύλλο. Θα πρέπει λοιπόν να διαμαρτυρηθούμε για οποιαδήποτε ε, επαναπατρισμό ή έκδοση, όπως έλεγε και η συνάδελφος Μπιόρκ. Ε, γνωρίζουμε πως επιστρέφονται γυναίκες σε χώρες από τις οποίες στις οποίες μάλλον χρησιμοποιήθηκαν ως εμπόρευμα θα ήθελα λοιπόν σε αυτή την έκθεση να αναφέρετε ρητά ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται να γίνεται. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, πυρογνώμονες και την ε, κυρία Χόνιμπολ που επιμένει και εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταίος από την κυρία ε, Γιούζο. Γιούτο, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Εγώ θα είμαι σύντομη γιατί διηγώθηκαν πολλά με τα οποία συμφωνώ. Σίγουρα από πλευρά μα στο εσωτερικό της έκθεσης, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το στοιχείο των ασφαλών ε, διαδρομών. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει στην αντιπροσωπεία μας και το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και σε άλλες εκθέσεις της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, είναι κάτι το οποίο πολύ πιστεύουμε και νομίζουμε πως είναι η μοναδική λύση που θα μπορέσει να εγγυηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα των όσων φεύγουν από καταστάσεις βασανιστήριων και πλήρους υποτίμησης της ανθρώπινης ζωής ε, όχι μόνο των γυναικών, είναι αυτό καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγγυηθεί την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων. Ήθελα να υπογραμμίσω και κάποιες στοιχείες που δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ή που αναφέρθηκαν ακροθυγώς. Το θέμα της ένταξης είναι κάτι που σίγουρα θα προσπαθήσω εγώ να εισάγω με τροπολογίες, ακριβώς ε, σε σχέση με τα όσα είπε η συγγήτρια Χάνιμπολ στην αρχή του σημερινής ακρόασης. Μετά από τις ε, ε, τρομοκρατικές επιθέσεις του Παρίσι υπήρξε μια τεράστια κλιμάκωση στις μορφές ε, ανοχής ε, και βία επεισόδια κυρίως κατά γυναικών που φορούν ε, το φουλάρι, την μαντήλα. Και αυτό γιατί οι γυναίκες σε αυτή την υπόθεση είναι πολύ πιο ευάλωτες. Σε σχέση με τον άντρα, η γυναίκα εύκολα μπορεί να αναγνωριστεί ακριβώς λόγω του διαφορετικού της φορέματος ή ενδύματος είναι λοιπόν ένα στοιχείο ε, διάκρισης που στην ουσία θα έπρεπε, ε, ε, που έρχεται μάλλον σε σύγκρουση με τη μεγαλύτερη ένταξη. Όλα τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη και που είχε και που θα έχει στο μέλλον προκύπτουν από το, οφείλονται μάλλον στο πρόβλημα της ένταξης και πάνω σε αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε. Να δούμε αυτό που συμβαίνει συχνά στις γυναίκες πρόσφυγες που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προθυμία τους να βγάλουν τα παραδοσιακά τους κοστούμια για να χρησιμοποιήσουν ε, συνήθειες και ήθη δυτικά, πολλές φορές αυτό παρεμποδίζεται από την ομάδα στην οποία ανήκουν, από την από τους ανθρώπους που τους συνοδεύουν, τους συντρόφους, την οικογένεια, την, την εθνότητά τους που ίσως να βρίσκονται και να ταξιδεύουν μαζί. Υπάρχουν δηλαδή φαινόμενα βίας απέναντι στις γυναίκες ε, που θέλουν ίσως να βγάλουν το φουλάρι, να αλλάξουν ζωή. Στην Ιταλία υπάρχουν ένα σωρό τέτοια επεισόδια έλλειψης ανοχής. Θα πρέπει λοιπόν ε, να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μικρά βήματα που οδηγούν προς την ένταξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να τους αναγκάσουμε να εγκαταλείψουν ε, τα ήθη και τα έθιμά τους, αλλά να τους αφήσουμε ελεύθερες. Πολύ συχνά δεν έχουν καν την ελευθερία να αποφασίσουν πώς θα ζήσουν, ε, πώς θα αντιθούν ακόμα και όταν θα φύγουν από τη χώρα προέλευσής τους. Ευχαριστώ. Thank you. That, that's η τελευταία σκιώδηση και πριν δώσω το λόγο στο επόμενο ναι, πρόσωπο να έρθω σε αυτό το θέμα της ένταξης αλλά δεν μιλούμε για αυτό μιλούμε για πρόσφυγες η ένταξη σημαίνει να τους βρει κανείς δουλειά να τους διευκολύνει να ενταχθούν να γίνουν μέρος δηλαδή του μέλλοντος του τόπου όπου διαλέγουν να μείνουν υπάρχουν χώρες μέλη όπου υπάρχει ε, μεγάλη ανοχή απέναντι σε ανθρώπους. Δεν γνωρίζω να υπάρχουν και μελέτες που να δείχνουν κάτι τέτοιο. Είναι το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο. Δεν είναι το πρόβλημα τόσο πολύ πώς ε, δίνονται οι άνθρωποι και τι εμφάνιση έχουν, Ο τους είναι αυτό. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ, τώρα ε, εσείς πρώτοι, και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαίρετη εκθεσή σας και αναφερόμενοι σε ορισμένα από τα θέματα που εξήγησαν οι προσκεκλημένες μας το πιο συγκλονιστικό είναι γυναίκες που γεννούν και όντας σε λοχεία συνεχίζουν το ταξίδι, συνεχίζουν την πορεία γιατί ανησυχούν ότι θα χάσουν την ευκαιρία να φτάσουν στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο το θέμα. Βεβαίως θα ήθελα να σας ρωτήσω να ε, δω τι σκέπτεστε. Βεβαίω και δεν θέλουμε να βάλουμε σε κέντρα κράτηση γυναίκε, ιδίω εγγύου γυναίκε ή που μόλι γέννησαν. Ούτε μπορούμε να παραβιάσουμε την θέληση μια γυναίκα που θέλει, προσπαθεί απεγνωσμένα να προχωρήσει, να φτάσει στη Γερμανία, σε κάποια άλλη χώρα τη Ευρώπη. Δεν ξέρω. Ήθελα λοιπόν ε, απαντήσει από εσά. γιατί είναι ένα από τα επίγοντα εκείνα ε, θέματα. Ο, ο χειμώνας έχει φτάσει. Ε, μας έχει έρθει. Πολλές από εμά που έχουμε και παιδιά ε, αντιλαμβανόμαστε πόσο τραγικό είναι το γεγονό αυτό. Όλο για τα κορίτσια, τα νεαρά κορίτσια που είναι τα πιο ευάλωτα θηλυκά όντα και δυστυχώς για όλα τα θέματα που μιλούμε από τη διακίνηση, από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την πορνεία, την γενετήσια κατάχρηση, ε, επίσης την ε, τον ε, γενετήσιο ακροτηριασμό των κοριτσιών κτλ. Όλα αυτά θίγουν κυρίως τα κορίτσια. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν ιδίω στόχευση σε αυτά τα παιδιά και για την διακίνηση. Εγώ θα το τόνιζα στην έκθεσή σας ακόμη περισσότερο. Έχουμε οδηγία για την διακίνηση και οι χώρες οφείλουν να την εφαρμόσουν. Πολλά από τα όσα συζητούμε εδώ έχουν σχέση με το γεγονός ότι δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι χώρες για να εφαρμόσουν, για να επιβάλλουν ε, τα μέτρα αυτά τα οποία είναι ήδη ε, ε, εγκεκριμένα και θεσπισμένα και συνεχίζεται μια τιμωρησία. Εξάλλου η μετεγκατάσταση είναι ηλεοφόρος για την είσοδό τους. Λίγες χιλιάδες έχουν μονάχα μετεγκατασταθεί σε άλλες ε, χώρες της Ευρώπης όπως έρχονται από την Τουρκία. Ειδικά για τις γυναίκες χρειάζονται νόμιμες διαδρομές. Για γυναίκες και κορίτσια θα ήταν και ο τρόπος να ξεφύγουν από όλη αυτή την βία στη βάση του φίλου το ζήτημα της κράτησης τώρα είναι πολύ σημαντικό να προστατευτούν τα παιδιά. Βάλαμε στο πακέτο του ασύλου το ζήτημα ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να κρατούνται ποτέ. Τα νεαρά κορίτσια λοιπόν δεν πρέπει να κρατούνται ποτέ. Γιατί είναι πρώτα παιδιά και μετά μετανάστριες. Και όντως ή άλλως το να είναι κανείς μετανάστης δεν είναι βάση για να κρατηθεί ως παιδί. Και το τελευταίο θέλω να τονίσω ένταξη, πρόσβαση στο σχολείο, ε, υπηρεσίας υγείας. Ένα τελευταίο αν με επιτρέπετε. Πήγα και είδα και την Λαμπεντούσα επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών ε, για την έκθεση της Σεσίλια Κένγκε. Ε, είδαμε το Ιταλικό ναυτικό, τα ίδια κάναμε και στο τουρκικό Μποντρούμ. Και θέλω να τονίσω τον εκπληκτικό ρόλο που έχουν αναλάβει οι μη κρατικές οργανώσεις αντιλαμβάνομαι τα όσα λέτε είναι αληθινά για τη χώρα για την οποία μιλήσατε και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι κανείς δεν μπορεί να επιστραφεί εκεί ε, κατ' εξαίρεση του κανονισμού του Δουβλίνου. Εγώ θέλω πάντως να αποτίσω φόρο τιμής στις μη κρατικές οργανώσεις. Είναι ιδιώτες, είναι οι γιατροί χωρίς σύνορα, είναι, αλλά και το, και το Ιταλικό ναυτικό που έχει φτιάξει ξεχωριστές εγκαταστάσεις υγείας για γυναίκες, για κορίτσια. Διεθνείς οργανισμοί όπως Safety for Children που έχουν φτιάξει μια διαδρομή για να παίρνουν παιδιά και γυναίκες από ε, τα σκάφη που έρχονται και να τα εντάσσουν σε ένα πρόγραμμα προστασίας. Ξαναλέω ευχαριστώ ιδιαίτερα το Ιταλικό Ναυτικό και στην Τουρκία, στο Μποντρούμ. Είδαμε και την παρουσία της ακτοφυλακής που συνεργαζόταν καλά με γυναική οργάνωση που λέγεται Καντήρ. Οι γυναίκες λοιπόν συνέρχονται και συνεργάζονται για να βοηθήσουν τις πρόσφυγες. Αυτά είναι λοιπόν θετικά παραδείγματα μιας έντονης κινητοποίησης της διεθνούς κοινότητας, της κοινότητας των μη κρατικών οργανώσεων, ιδίως για ζητήματα δηλαδή προσφύγων, ασύλου και αυτό ήθελα πολύ να το τονίσω. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλη εγγεγραμμένη. Α, εσείς Τζούλη. Δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο. Και μένα με έχει συνεπάρει συναισθηματικά η συζήτηση αυτή και οι παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων και θετικά και βεβαίως πολύ αρνητικά συναισθήματα αισθάνομαι. Είναι πραγματικά ε, συγκλονιστικό να ακούει κανείς τις ιστορίες αυτές που διηγείστε και ω γυναίκα βέβαια με παιδιά. Πολύ δύσκολο να τα ακούω αυτά. Άκουσα βέβαια και ε, πολύ θετικά πράγματα. Αναφέρομαι στην Γιάλα Τράπαν και εγώ έχω ένα ιστορικό συμμετοχή σε κοινωνική οργάνωση στην ε, Βόρειο-Δυτική Αγγλία όπου έχουμε, είχαμε και έχουμε τη θέληση να ε, στήσουμε στα πόδια τους εναλλακτικά οικονομικά συστήματα που να προσφέρουν κάποια ελπίδα στον κόσμο και συχνά πρόκειται για κοινότητες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ε, σημαντικές προκλήσεις και βλέπουμε ότι εκείνοι οι άνθρωποι έχουν εντονότερο και, το, ε, και την επιθυμία του να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Εξακολουθώ ωστόσο να είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη για το ζήτημα της κράτησης και θα ήθελα να ρωτήσω τι σκέπτεται σχετικά με την ανακοίνωση του Τούσκ που λέει ότι θα πρέπει να κρατούνται οι πρόσφυγες για ένα 18 μήνο και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στα πιο ευάλωτα από τα πρόσωπα αυτά για τα οποία μιλούμε τώρα δηλαδή γυναίκες και νεαρά κορίτσια ή παιδιά. Άλλος βουλευτής που θέλει να λέει το λόγο, παρακαλώ. Ωραία. Κανείς. Οπότε, οι προγνώμονες ε, αρχίζονται σαν Η Χριστίνα. Πέντε λεπτά το πολύ, παρακαλώ. Νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω σου ειδικά. Δεν είχα προετοιμαστεί, αλλά άκουσα πολύ προσεκτικά τις τρεις συναδέλφους. Είμαι εντυπωσιασμένη από το έργο τους και από αυτά που μας είπατε. Σήμερα ο κόσμος μας είναι χαοτικός για ποικιλία λόγων. Αν όμως ανατρέξουμε στην ιστορία, συνειδητοποιούμε ότι οι γυναίκες και τα παιδιά την πληρώνουν τις περισσότερες φορές, ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσεων. Το ελάχιστο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάστασή τους. Έστω και μια πολύ μικρή βελτίωση έχει σημαντικά απτά αποτελέσματα στην πράξη. Άκουσα σήμερα για τις προτάσεις στην έκθεση της κυρίας Χάνιμπολ και συνειδητοποιώ ότι αν καταφέρουμε να ενσωματώσουμε και κάποιες προτάσεις, και συστάσεις, το κέρδος θα είναι μεγάλο. Ο χρόνος πιέζει πάντως. Σήμερα το θέμα δεν είναι να φτάσει κανείς δεν αρκεί να φτάσει κανεί σε μια χώρα για να λύσει το πρόβλημά του, για να είναι προστατευμένος. Όπου και αν ζει κανεί στην Ευρώπη, σήμερα, έχει ανάγκη υποστήριξη, συνεργασία. Χρειάζεται η κοινωνία των πολιτών και το εκάστοτε δημόσιο να συνεργαστούν. Και οι δημόσιο τομέα μαζί με την ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει επίση να συνεργαστούν να εξεύρουν νέους τρόπους σύμπραξης. Στη Σουηδία αυτό κάναμε. Προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε τουλάχιστον τον ενθουσιασμό που υπάρχει στη βάση. Ελπίζω ότι οι βελτιώσεις που θέλετε να επιφέρετε θα γίνουν πραγματικότητα το συντομότερο δυνατόν. Πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις πρέπει να τύχουν τις ε, ολοθερμής υποστήριξης μας. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Η Ντέπορα. Με φορμή προηγούμενα σχόλια σχετικά με τη διαδικασία χορηγήσης ασύλου τις λεγόμενες ασφαλείς χώρες ε, και το θέμα της κράτησης. Λοιπόν, σχετικά με τις ασφαλείς χώρες είπαμε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τη διαδικασία. Είπαμε ότι χρειάζεται να ληφθεί υπόψη το φύλλο. Και να δούμε αν πραγματικά ο κατάλογος των ασφαλών χωρών ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα αυτό εξαρτάται, το κατά πόσο δηλαδή είναι ασφαλής μια χώρα ή όχι, εξαρτάται από το αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Ίσως να χρειάζονται δύο ξεχωριστοί κατάλογοι, γιατί κάποιες ε, χώρε μπορεί να είναι ασφαλεί για του άνθρωπους αλλά όχι για τις γυναίκες. Ίσως και το αντίθετο σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό ε, ανεξαρτήτω του κατά πόσο υπάρχουν πραγματικά ασφαλείς χώρε. Πάντω, θετικός κατάλογος ασφαλών χωρών σημαίνει ότι μπορεί να επαναπροωθεί πολύ εύκολα με σχετικά συνοπτικές διαδικασίες. Μετά από συνοπτική δηλαδή σύντομη κράτηση. Οπότε είναι πολύ ε, σχετικός ο θετικός κατάλογος ασφαλών χωρών για τις Τώρα για το θέμα της κράτησης. Πιστεύω ότι η κράτηση είναι κακό πράγμα. Για όλους. Για οποιονδήποτε. Όταν μιλάμε για άσυλο, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν υποστεί τραυματισμό, ψυχικά τραυματισμένους. Σε πως κανείς ετών άσυλο δεν πρέπει να κρατείται. Αυτό θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα στισμένη αποτελέσματα σε ευάλωτες ομάδες, κυρίως παιδιά που βεβαίως δεν πρέπει ποτέ να κρατούνται, σε γυναίκες, εγγύους, θύματα βίας, Γνωρίζουμε από μελέτες ότι η κράτηση στις ευάλωτες αυτές ομάδες προκαλεί επιπλέον ψυχικό τραυματισμό ανεξαρτήτως τη διάρκεια της κράτησης. Και τέλος, συζητήσαμε το θέμα της εφαρμογής στην πράξη συγκεκριμένων καλών πολιτικών που δυστυχώς όμως δεν εφαρμόζονται. Τα κράτη-μέλη δηλαδή δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να τις υλοποιήσουν στην πράξη. Το είπαν πολύ αυτό. Γνωρίζω πολύ καλά ότι κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει γυναίκες να τους χορηγηθεί άσυλο γρήγορα με την πρώτη και να μην υποστούν όλα τα προβλήματα είναι η αξιοπιστία του συστήματος αξιολόγησης. Μίλησα με 100 γυναίκες ετούσες και σε όλες τις περιπτώσεις μας είπαν ότι έχουν αμφιβολίες την αξιοπιστία του συστήματος. Αυτές τώρα μας βοηθούν και έτσι ακούγεται περισσότερο και η φωνή των γυναικών στη διαδικασία αυτή. Υποστηρίζουμε επίση τη σχετική εκστρατεία και αυτό νομίζω πρέπει να το προσθέσουμε στην έκθεση. Ε, πρέπει να είναι μία από τι συστάσεις μας, δηλαδή μέτρα για την αξιοπιστία του σύστηματος αξιολόγηση των αιτήσεων. Υπάρχουν πολλά πρακτικά πράγματα που μπορούν να γίνουν προ την κατεύθυνση αυτή για να υπερπηρήσουμε και το θέμα τη έλλειψη εμπιστοσύνη την δυσπιστία απέναντι στο σύστημα, κυρίως από την πλευρά των γυναικών που αιτούνται άσυλο. Πρόεδρος. Και τώρα η Ανδρέα. Μια που πηγαίνουμε ανάποδα. Ευχαριστώ. Να έρθω στο θέμα τη συνέχιση της πορείας των γυναικών και η κυρία Ρέιλι ίσως πει περισσότερα από την άποψη του είπα του αρμοστή των Ηνωμένων αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ουδέτερου χαρακτήρα πληροφορίε στους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμα σε πορεία για το ποιε είναι οι επιλογές αν δεν περάσουν από τα hotspot αλλά και ποιε είναι οι υπηρεσίε στι οποίες μπορούν να αναφερθούν. Και εδώ έχουμε βέβαια απέναντί μας τις ε, πληροφορίε των διακινητών και ανθρώπου που έχουν επενδύσει στο ταξίδι αυτό και θέλουν να συνεχίσουν. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για του οποίου οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να συνεχίσουν την πορεία. Συχνά οι άνθρωποι δεν έχουν καν υπόψη, δεν έχουν ιδέα για τι συνθήκε που επικρατούν στι χώρε προορισμού αλλά και στι χώρε μέσα από τι οποίε θα περάσουν. Και προσπαθούμε να χαρτογραφήσουμε τι ε, συνθήκε αυτέ, ώστε να γνωρίζουν οι ενδεχόμενοι πρόσφυγες ποιε θα είναι οι καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν και στις χώρες με την κατάσταση και στις χώρες μέσα από τις οποίες θα περάσουν ή σε αυτές που θα αποφασίσουν να μείνουν. Εδώ ε, χρειάζεται και κάποια προσοχή για του ανθρώπου αυτού που ορισμένοι λένε ότι είναι η μεγάλη πορεία. Το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο όπου επιθυμούν. Και το θέμα που ανέφερε και η κυρία Μπίλτ τη μη επιστροφή που εφαρμόζεται τώρα για την Ελλάδα ε, εκτός, ε, ε, εκτός κανονισμού Δουβλίνου. Είναι δύσκολο να πείτε στους ανθρώπους ότι πρέπει να παραμείνουν εκεί, να σταματήσουν εκεί, γιατί οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Βέβαια, αν ζητήσουν περισσότερη άσυλο το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να αντιδράσει. Αν περισσότεροι ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα θα μπορεί το σύστημα να ανταποκριθεί. Ένα άλλο θέμα για την μετεγκατάσταση που εμείς βλέπουμε σαν μια νόμιμη οδό. Ε, υπάρχει ποσόστος 22.000 που πρέπει να επανεξεταστεί και θα πρέπει να είναι προβλέψιμο πόσοι φτάνουν στην επικράτεια μιας συγκεκριμένης χώρας μέλους. και δύο λόγια για την ανακοίνωση του Ντόναλτ Τούσκ. Διάβασα σύντομα ένα άρθρο σήμερα το πρωί. Νομίζω ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει μια σύγχυση στα κεφάλια ορισμένων σχετικά με το ποιος είναι μετανάστης και ποιος είναι πρόσφυγας. Μιλούσε για 18 μήνες. Υπάρχει όμως η οδηγία που λέει ότι μόνο υπό ειδικέ, υπό έκτακτες ε, συνθήκες μπορεί να κρατηθεί κάποιος μέχρι 18 μήνες και αυτές πρέπει να έχουν επιβληθεί από δικαστήριο. Νομίζω ότι ο Τούσκ δεν μιλεί για ανθρώπους που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας. Αν δεν μιλεί για τους ανθρώπους αυτούς, ή πάνω, αν μιλεί για τους ανθρώπους αυτούς, τότε σημαίνει ότι παραβιάζει τις συνθήκες, αλλά και την οδηγία, το άρθρο 8 και 9 της οδηγίας που λέει ότι χρειάζεται σύντομη διεκπαιρέωση δυνατόν ε, ε, ε, συντομότατη κράτηση και ούτω καθεξής. Θα περιοριστώ σε αυτά. Ευχαριστώ. Τέλος η Ναι. Όλες οι συστάσεις μας τρεφονται γύρω από την προστασία γυναικών και κοριτσιών όταν βρίσκονται εν κινήσει δεν είναι κλασική η περίπτωση ανθρώπων που είναι εγκατεστημένοι κάπου και μπορούν να τους βρουν θέση με προγράμματα πολυτομιακά κλπ. Όλα όσα είπα για καλύτερη διαμεθοριακή ε, συντονιστική προσπάθεια για την διαβίβαση πληροφοριών, για συντονισμό ε, των απαντήσεων. Επίσης κοινά κριτήρια του ευάλωτου. Εφόσον περνούν από μια χώρα σε άλλη, οι αρχές να μπορούν να εντοπίζουν αμέσως ποιες ομάδες ανθρώπων είναι οι πιο ευάλωτες. Να τους εντοπίζουν και να τους προσφέρουν χέρι βοήθειας. Και βεβαίως χρειάζεται και μια καινοτόμα προσέγγιση στο πώς θα κάνει κανείς εργασία πρόληψης των ε, ε, ενδεχόμενων γενετήσεων επιθέσεων, βιασμών κ.ο.κ. Επίσης διάθεση προφυλακτικών, εκεί που θα χρειαστούν αυτά τα πράγματα όλα. όχι στα νοσοκομεία. Σε ό,τι αφορά τη στόχευση στις ομάδες των κοριτσιών, η έρευνά μας δείχνει ότι η ομάδα που ε, περνά τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι τα κορίτσια και ιδίως κορίτσια που κινούνται μόνα τους ή είναι απομονωμένα όταν αναγκάζονται να αναλάβουν πολύ νωρίς ε, ρόλους ενηλίκων, είτε για την προστασία μικρών αδελφών, είτε και ως ανήπικες μητέρε, τότε είναι πάρα πάρα πολύ ευάλωτα τα παιδιά αυτά. Έχουμε κάνει πολλέ έρευνε και παγκόσμια δηλαδή για τα πράγματα αυτά και για το ότι πρέπει να εντοπίζονται τα ανήλικα κορίτσια γιατί είναι και οι πιο ε, κρυφές ομάδες, πιο κρυμμένες ομάδες μέσα στους πληθυσμούς αυτούς. Αναγνωρίσατε εσείς προηγουμένως την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι μικρατικές οργανώσεις. Ε, δέχομαι ευχαριστώ το σχολείο σας αυτό. Όπως είπα, ήταν μια αποστολή αυτή που, στην οποία συμπράξαμε των Ηνωμένων Εθνών. Η επόμενη αποστολή μας θα είναι πάλι ε, Βοσνία, Σερβία και Σουηδία και θα ε, εργαστούμε με γυναίκες τις, με, με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχει διαφορά με την Ιταλία όπου είναι πιο εγκατεστημένος ο πληθυσμός. Δεν είναι τόσο πολλοί ομάδες που κινούνται με τέτοια ταχύτητα όπως μέσω Ελλάδας και μέσω των Βαλκανίων. Ίσως λοιπόν εκεί δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω. Ίσως το πλαίσιο εκεί να είναι καλύτερο. Ναι βεβαίως υπάρχει πεντούσα σωστά. Πάντως ε, σημειώνω το σχόλιο σας για την συμβολή των ε, ε, οργανώσεων των ισχυρών των πολιτών όμως και στην Ελλάδα και στη Μακεδονία είδαμε, είδαμε τα σημαντικά προβλήματα. Αν και στα ελληνικά νησιά δεν είδαμε ε, γυναικείες ομάδες, δεν είδαμε καν ε, οργανώσεις μικιό δηλαδή. Πάντως το επόμενο, η επόμενη προσπάθειά μας θα να συνεργαστούμε με τις οργανώσεις αυτές. Ναι. Η κυρία Μπάλ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ δύο στις εμπειρογνώμονες. Εγώ πάντως έμαθα πολλά πράγματα σήμερα και τη σπουδαία δουλειά που κάνετε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για τα λόγια που μας είπατε. Λίγες παρατηρήσεις τώρα, καθώς κλείνω. Τα όσα κάνουμε και εμείς, τα όσα κάνουν βεβαίω και οι μυρογνώμονες εδώ και πολύ καιρό και, και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι να φέρουμε σε φως πράγματα που συμβαίνουν και που δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί. Και ιδίως για την βίας τη βάση του φύλου, ιδίω σε βάρος γυναικών και παιδιών και όλο αυτό το θέμα της γενετήσιας βίας σε βάρος γυναικών προσφύγων πραγματικά ε, έχει τρομακτικές διαστάσεις και ακούσαμε ε, πραγματικά σε βάθος πράγματα θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε γνωστό το πρόβλημα όχι μονάχα οι άνθρωποι που γνωρίζουν πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο γιατί πρόκειται για ένα από τα ζητήματα κλειδιά. Πρέπει να αναγνωριστεί και όσο είναι δυνατόν να προληφθεί. Και όλη αυτή η ιστορία της αξιοπιστίας που συνδέεται με αυτό όταν οι γυναίκες έρχονται στα κέντρα υποδοχής και ζητούν άσυλο και δεν τις πιστεύουν οι αρμόδιοι. Βεβαίω μπορεί να μην υπάρχουν ενδείξεις μπορεί να είναι δύσκολο για αυτέ να μιλήσουν για τα όσα του έχουν συμβεί. Όλα αυτά πρέπει να μας απασχολήσουν περισσότερο και η ευαισθητοποίηση όπου μπορούμε διότι βέβαια εάν υπάρχει δυσπιστία ε, στην φάση της υποδοχής οι επιλογές είναι τρομακτικές ή πάει κανείς στο δικαστήριο που ε, και υπό καλές συνθήκες θα προτιμούσαν να το αποφύγουν ή δεν λαμβάνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και είτε μπαίνουν σε κράτηση είτε επιστρέφονται. Χρειάζεται λοιπόν να συζητήσουμε, συζητήσαμε άλλωστε εκτεταμένα σήμερα το ζήτημα της προστασίας των γυναικών, μιλήσαμε γι' αυτό, ιδίω βέβαια για τα κορίτσια που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερου κινδύνου, αλλά και οι γυναίκε γενικότερα χρειάζονται ασφαλείς διαδρομέ. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση για το πόσο επικίνδυνα τα πράγματα. Άκουσα με ενδιαφέρον πριν τη συζήτηση για το θέμα ότι οι πρόσφυγες και ειδικότερα οι γυναίκες θέλουν να παραμείνουν ανώνυμες, δεν θέλουν οι άλλοι να ξέρουν ποιες είναι. Έχουν αυτή την επιθυμία να μην, να μην γίνουν γνωστές οι περιπτώσεις τους, κάτι το οποίο βέβαια καθιστά δυσκολότερη ακόμη την προστασία. Προφανώς μόνο υπό ακραίες περιστάσεις ε, δεν ε, θέλει κανείς να γίνει γνωστή η περίπτωσή του. Έχουμε λοιπόν πολλά πράγματα. Και το ερώτημα είναι και το ερώτημα τι γίνεται να φτάσουν στον τόπο προορισμού και τι κάνουν όταν φτάσουν εκεί και αυτό το project για άλλα πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η έκθεση κάνει την προσπάθεια να παρακολουθήσει την διαδικασία από την αρχή, από το ξεκίνημα της πορείας της πρόσφυγος μέχρι την άφηξή της στο τελικό προορισμό και την προσπάθεια να στήσει μια ζωή εκεί. Εγώ από την σκοπιά μου ως εισηγητρίας βρήκα πολύ χρήσιμη την ακρόαση. Πολλά από αυτά λοιπόν θα τα περιλάβω. Είμαι βεβαίω ότι θα δεχθώ και πολλές τροπολογίες σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι όλες για τα όσα μας παρουσιάσατε. Um, Λίγη τώρα η ακρόαση. Έχουμε δυστυχώς ακόμη ένα θέμα στην ημερησία διάταξη της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών. Όσοι εξημών ήρθατε ειδικά για την ακρόαση και επιθυμείτε να αποχωρήσετε, δύναστε να το πράξετε. Οι ευρωβουλευτές σας παραμείνουν γιατί έχουμε ένα τελευταίο θέμα. Μείνετε λοιπόν για λίγα λεπτά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 Μπορούμε σύντομα να διεκπαιρεώσουμε και το τελευταίο σημείο της ημερήσιας. Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Γκρέκνερ είναι η συγγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μέρη για όλες ακόμη που κρατούν εδώ τα μετερίζια σε αυτή την προχωρημένη ώρα θα προσπαθήσω εν συντομία να εξηγήσω τη γνωμοδότηση για ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο θα είχε κανείς πολλά να πει. Βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι είναι περασμένη ώρα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομη. Πρόκειται για το μισθολογικό dumping και τον αγώνα κατά του μισθολογικού dumping. Εδώ βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Πού να αρχίσω από πού να αρχίσω να σας τα εξηγώ. Θα προσπαθήσω να τονίσω ορισμένες πτυχές που είναι σημαντικές και ειδικότερα για εμάς τις γυναίκες. Αυτό το ε, ε, μισολογικό ντάμπινγκ έχει πολύ σχέση και με τους αποσπασμένους εργαζόμενους, αλλά πηγαίνει και πολύ μακρύτερα από αυτό, διότι η ε, σημαντικότερη συνέπεια του ε, μισολογικού ντάμπινγκ είναι ε, η μαύρη εργασία. Εκεί χρειάζεται αντίδραση και αντιμετώπιση. Αυτό το μισολογικό ντάμπινγκ γίνεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Όταν κάποιος είναι υποχρεωμένος για να επιβιώσει, να δεχτεί οτιδήποτε, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, οι δίθεν ανεξάρτητοι, αυτούς χτυπάει περισσότερο. Και είναι πραγματικά λυπηρό. Μπορεί να πάρει λοιπόν διάφορες μορφές το μισθολογικό ντάμπινγκ. Και μάλιστα σε ορισμένους κλάδους είναι εντονότερο. Εδώ χρειάζεται να γίνουν ορισμένα πράγματα. Θα τονίσω ορισμένους κλάδους που πλήττονται βαριά από το μισθολογικό ντάμπινγκ και ιδίως βέβαια για τις ε, γυναίκες αφενός ο κλάδος των οικιακών βοηθών νοσηλευτριών στο σπίτι εδώ γίνονται πάρα πολλά κρυφά εδώ θα περιλάβω και ορισμένα από την έκθεση για τις ιατρικές βοηθούς. Αυτά πρέπει να διασυνδεθούν εδώ γιατί εκεί γίνονται πολύ καλές προτάσεις στην έκθεση αυτή που εννοώ. Συχνά πρόκειται για γυναίκες οι οποίες αναγκάζονται να αφήσουν τις οικογένειές τους σε άλλη χώρα για ένα ε, χρονικό διάστημα για να μπορούν να ε, προσφέρουν τις ε, υπηρεσίες αυτές, νοσηλευτικές και άλλες, και επιστρέφουν μετά όταν μπορούν στις ε, χώρες τους και στις οικογένειές τους. Μεγαλώνουν τα παιδιά χωρίς μητέρα, ε, χωρίζουν ε, οι οικογένειες, λείπουν οι γυναίκες από πολλές χώρες. Έχουμε βέβαια και άλλους κλάδους που είναι κλασική κλάδοι απόσπασης εργαζομένων όπου αν εξετάσουμε θα δούμε και εκεί να, να πλήττονται πολλοί γυναίκες. Παράδειγμα, όπου υπάρχουν πραγματικά τρομακτικές περιπτώσεις κοινωνικού και μισθολογικού ντάμπινγκ, κυρίως ο τομέας της μεταποίησης του κρέατος. Τον φέρνω ως παράδειγμα και για άλλους τομείς, όπου μπόρεσα κρυφά να παρακολουθήσω τι ε, συμβαίνει. Γυναίκες που ε, κρυμμένες σε κάποια πίσω δωμάτια τεμαχίζουν κοτόπουλα και ε, τα συσκευάζουν υπό άθλιες συνθήκες. Έχω και το άλλο παράδειγμα της Ryan Air με... που θα έπρεπε και εκεί να εγγύψουμε περισσότερο στο τι συμβαίνει. Νομίζω ότι το τμήμα της περιγραφής της καταστάσεως δεν θα πρέπει να είναι πολύ μακρό, διότι βεβαίως μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και όλες γνωρίζουμε περιπτώσεις. Από την άποψη της ε, Επιτροπής μας πρέπει να γίνουν κάποιες πρακτικές προτάσεις, πρακτικές συστάσεις. Εγώ έχω δει εδώ ένα, μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόσπαση εργαζομένων που είναι του Σεπτεμβρίου 2014 και έχουμε ακόμα επίκαιρη. Δεν υπάρχουν εδώ ωστόσο, δεν περιλαμβάνει στατιστικές για γυναίκες, τουλάχιστον όχι πολύ χρήσιμες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ειδικά στους τομείς εκείνους όπου γνωρίζουμε ότι σημειώνονται πολλά προβλήματα Χρειαζόμαστε πιο γλαφυρές στατιστικές, πιο ξεκάθαρες στατιστικές και να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει κλάδους και να εντοπίσει κλάδους όπου και εντός των κλάδων δηλαδή που ε, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις γυναίκες και όπου εκεί σημειώνεται μισθολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ. Μπορεί να διασυνδεθεί η ιστορία αυτή και με την μαύρη εργασία. Βεβαίως, να γίνει η διασύνδεση αυτή πάντοτε υπό την ειδικότερη οπτική γωνία των γυναικών. Και για να συνεχίσω με τις πρακτικές συστάσεις, νομίζω ότι είναι ε, σημαντικό και θα είναι σημαντικό να υπάρξει ένα δίκτυο που να εξετάζει τις ιστοσελίδες. Υπάρχει και μια θαυμάσια ιστοσελίδα που δίνει πληροφορίες για τις αποσπάσεις εργαζομένων στον κλάδο της οικοδομής. Πρέπει λοιπόν να στρέψουμε τα βλέμματά μας πάλι, ξαναδέω στους κλάδους εκείνους όπου ε, ενδιαφέρουν περισσότερο τις γυναίκες. Μπορούμε και εδώ να κάνουμε μια προσπάθεια. Είδα και εδώ στην έκθεση της κυρίας Κούνεβα την οποία προανέφερα ότι υπάρχουν πληροφορίες και μπορούμε να αποκαταστήσουμε ένα σύνδεσμο με αυτό το περιεχόμενο σε αυτής της εκθέσεως. Στην Αυστρία υπάρχουν παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ Ουγγαρίας και Αυστρίας όπου άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι απαιτήσει που έχουν απέναντι στον εργοδότη και ούτω καθεξής μπορούν να προσφύγουν σε ένα γραφείο. Ε, αυτό λειτουργεί τόσο καλά, διαδίδεται ε, η διεύθυνση του γραφείου, το αριθμό τηλεφώνου κτλ. ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να προσφέρουν σε αυτό. Πρόκειται για βασικέ πληροφορίε και να γνωρίζουν ότι να, εδώ υπάρχει ένα συνομιλητή και μπορώ να του μιλήσω και μπορώ να λάβω υποστήριξη από αυτόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό στην γνωμοδότηση δίνω ιδιαίτερο βάρο σε αυτέ τι πρακτικέ συστάσει. Τέλος, τονίζω μια ακόμα πρακτική σκοπιά, το ζήτημα της ευθύνης και του υπεργολάβου, για παράδειγμα που ε, έχουν ε, εργαζόμενες μερικής απασχόλησης για οικιακές υπηρεσίες κλπ. και που εκεί ε, φροντίζουν να αποφεύγουν όσο είναι δυνατόν την εφαρμογή των νόμων, να φροντίσουμε ώστε να αποφεύγεται το μισθολογικό ντάμπινγκ και το κοινωνικό ντάμπινγκ όσο γίνεται περισσότερο και αυτό κυρίως που ε, πλήττει τις γυναίκες. Ευχαριστώ, Εύελεν. Η ε, Μικαέλα θα ήθελα να πάρει το λόγο. Θέλει κάποιος άλλος? Όχι, ωραία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία, την ησυχήτρια που παρουσίασε αυτήν την ε, γνωμοδότηση. Κατά τη γνώμη μου, τα μέτρα που προτείνεται είναι πολύ πρακτικά για να μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό dumping εναντίον των γυναικών. Ε, δεν ξέρω αν είναι απόλυτη αρμοδιότητα δική μας. Ε, βασικά είναι αρμοδιότητα της ε, ΕΜΠΛΕ, της Επιτροπής Απασχόλησης. Εγώ θεωρώ πως είναι ένα ζήτημα, ωστόσο, που έχει να κάνει με τον αθέμητο ανταγωνισμό. Πρέπει να το καταπολεμήσουμε λοιπόν, να καταπολεμήσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά και αυτοί που το αντιμετωπίζουν πρέπει να το καταπολεμήσουν, δηλαδή οι ε, εργαζόμενοι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση και είναι το σημείο 2 και 3 στη δική σας νομοδότηση και αυτά είναι αυτά που αφορούν τις πληροφορίες, ε, ε, τη δυνατότητα μάλλον να ενημερώνονται όσο γίνεται περισσότερο οι ε, εργαζόμενοι. ώστε να μπορούν οι ίδιοι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους έναντι αυτών των πρακτικών. Όταν είναι ενήμεροι μπορούν να προβούν στη λήψη των σωστών αποφάσεων και νομίζω πως αυτό είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Στηρίζω λοιπόν τα σημεία 2 και 3. Δεύτερο τώρα ε, μέσο που θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό και το κοινωνικό dumping είναι μια σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας που ήδη ισχύει σήμερα, δηλαδή την οδηγία για τις υπηρεσίες και την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Νομίζω πως θα αναφέρετε στην γνωμοδότησή σας, όμως έχω ένα προβληματάκι με αυτό και εδώ έχω είναι η ομαύρη λίστα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αυτό διότι Αυτό σημαίνει ότι στιγματίζουμε συγκεκριμένους εργοδότες. Είναι πολύ, νομίζω, σκληρό το οποίο μπορεί να είναι κατάλληλο σε περίπτωση εγκληματικής δραστηριότητας ή σε περίπτωση που τίθεται η ζωή κάποιου σε κίνδυνο, αλλά δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο εργαλείο σε αυτή την περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την πρότασή της. Πιστεύω πως θα, με, θα είναι επιτυχής αυτή η γνωμοδότηση και θα καταθέσουμε και τροπολογίες. Ευχαριστώ. Για να κλείσουμε ανακεφαλαιώνοντας. Ναι. Πολύ γρήγορα. Κυρία Ρέγνη, σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και για τις προτάσεις σας. Ευχαρίστω τα δέχομαι. Ε, θα έχουμε ασφαλώς ευκαιρία να συνεργαστούμε και με τις άλλες και όλες τις και να διεξέλθουμε τα διάφορα θέματα. Μία σύντομη παρατήρηση μόνο για τον μαύρο κατάλογο των εργοδοτών. Έχω να σου πω το εξή. Είμαι και μέλος στην Επιτροπή Τάξε και εκεί είδαμε όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα με την ε, φοροδιαφυγή με την επιθετική αυτή φόρο αποφυγή, με τα Starbucks και McDonald's και όλα αυτά τα σχετικά. Καμιά φορά είναι αναγκαίο να κατονομάζονται οι επιχειρήσεις, γιατί στις περιπτώσεις αυτές αντιδρούν μόνον όταν κατονομαστούν. Θα χρειαστεί να μιλήσουμε για αυτή την μαύρη λίστα δεν ε, εννοώ βεβαίω ότι θα πιάσουμε την κάθε μικρομεσαία επιχείρηση που κάποια στιγμή πέπεσε σε ένα σφάλμα. Αλλά όταν ε, υπάρχει συστηματικά ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στο dumping, αυτό θα πρέπει να ε, καταδειχτεί, να κατονομαστεί και θα δούμε με ποιο τρόπο είναι πιο αποτελεσματικό να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Πριν κλείσουμε. Δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα. μία υποβολή τροπολογιών 16 Δεκεμβρίου. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου. Ψηφι... Ψηφίζουμε την έκθεση στην ΕΜΠΛ 22 Μαρτίου και πάμε στη Ολομέλεια του Απριλίου πλέον για την Ολομέλεια, για την ψηφορία στην Ολομέλεια. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που μείνετε τόσο αργά. Πέμπτη. Πέρα συνδυάσεως.